colleagues, Συνάδελφοι, ας ξεκινήσουμε λοιπόν ξανά. Καταρχήν να σας ε, ε, παρουσιάσω τα αποτελέσματα της συνάντησης των συντονιστών. Ξέρω ότι όλα αυτά είναι πολύ επαναλαμβανόμενα, αλλά πρέπει να το κάνω. Οπότε προσδεθείτε και ακούστε Όλα τα αιτήματα για την συναντήση του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου ελήφθησαν υπόψη. Η διαδικασία του κατεπήγοντος θα εφαρμοστεί στην 960 για την ε, δημιουργία του εμπορικού κέντρου στο Μιλάνο. Η αιτήσια έκθεση του 2018 Ήδη είχε ληφθεί απόφαση με γραπτή διαδικασία, οι συντονιστέ την επιβεβαίωσαν. Προγραμματισμό για του επόμενου μήνε. Έλειψαν υπόψη όλα τα αιτήματα. Οι συντονιστέ αποφάσισαν ότι οι αποφάσει όμω θα ληφθούν αργότερα, κατά τη διάρκεια τη συνήθου διαδικασία. Ζητήθηκε από τη Γραμματεία να καταγράψει όλες τις αναφορές και να τις υποβάλει στην επόμενη συνάντηση έτσι ώστε να συζητηθεί και το θέμα ενός ενδεχόμενου μπαλεγιάς ξεκαθαρίσματος. Σε ό,τι αφορά τις συστάσεις, τις αμφισβητούμενες συστάσεις για την 757 ε, και 754 και 755 ε, ε, ψηφίστηκε όπως είχα ζητήσει εγώ ε, η 426 ε, έκλεισε, η 454 και 456 ε, όπως ζήτησαν οι ε, πράσινοι. Στην, στις επισκέψεις μας και τις ακροάσεις μας ε, λάβαμε γνώση τους, την καινούργια λίστα για τους συμμετέχοντες στη Βαλετόρα Ε, και με την Εύη και την Ήτρε συμφωνήσαμε μια μία κρόση για την ε, άρνηση της κλιματικής αλλαγής. Για το πρόγραμμα του ε, Ελληνικού Συνεδρίου για το 2020 συνεισφορές μέχρι τις 6 Ιανουαρίου μετά το ΕΛΚ στα διάφορα μας ενημέρωσε ότι επιθυμεί να διοργανωθεί μια επίσκεψη στη χώρα των Βάσκων μετά τις ε, εκλογές της αναφοράς 15-25. Καλωσορίζουμε την Λίνα Βοσιλιούτε και την Τζένιφερ Αλσόπ. για να μας παρουσιάσει, παρουσιάσουν την επικαιροποίηση της μελέτης είναι κατάλληλη για το σκοπό αυτό η οδηγία για την υποβάθμιση και η ποινικοποίηση της ανθρωπιστικής βοήθειας στους παράτυπους μετανάστες. Θα σας δώσω το λόγο για 20 λεπτά. Έχετε νομίζω και μια παρουσίαση έτσι δεν είναι. Να, ωραία, τη βλέπουμε. Ευχαριστώ πολύ την ε, Επιτροπή σας ε, που μας ανέθεσε αυτή τη μελέτη. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Είδαμε ότι η ποινικοποίηση της αλληλεγγύης δεν έχει εμφανιστεί σε ένα πολιτικό και νομικό κενό. Υπάρχουν συγκυριακοί παράγοντες που οδήγησαν σε αυτή την ποινικοποίηση της αλληλεγγύης ε, προς ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια, παράτυπους μετανάστες και πρόσφυγες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένας από τους παράγοντες είναι ότι η εθνική και κοινωνική νόμη δεν είναι σαφή ό,τι αφορά το λαθρεμπόριο μεταναστών και τον ορισμό του. Δεύτερον, ο αγώνας για, εναντίον της, του λαθρεμπορίου μεταναστών ε, έχει εμπλακεί με την ποινική δικαιοσύνη, με το στρατό, με τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών κλπ. Οπότε δεν είναι σαφές το τι κάνουμε και για ποιο λόγο κάθε φορά. Αν η, ε, το λαθρεμπόριο μεταναστών είναι έγκλημα, θα πρέπει να οριστεί καλύτερα στο ποινικό δίκαιο. Τρίτον, η μονομερής δράση και η έλλειψη ε, λύσεων και αλληλεγγύη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Βλέπουμε ότι ε, πολλοί θέλουν να μετακινήσουν ευθύνε σε άλλα κράτη-μέλη ή στην κοινωνία των πολιτών εξαιτία τη αδυναμία του να λύσουν μακροπρόθεσμα τα προβλήματα τη μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε γίνονται από δύο πομπέι τράγοι ή εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών πολλές φορές. Να δούμε έναν έναν από τους παράγοντες. Πρώτος παράγοντας, όπως είπαμε, η νομική ασάφεια. Να δούμε σε βάθος τι είναι και τι δεν είναι παράνομο. Όπως βλέπετε το άρθρο 1 τη οδηγία 2002 λέει ότι οποιοδήποτε άτομο που εκουσίω βοηθάει ένα άτομο που δεν είναι ε, πολίτης της ε, κράτους μέλους να μπει ε, να εισέλθει στην επικράτεια το, του κράτους μέλους κατά παράβαση των νόμων του κράτους μπορεί να κατηγορηθεί για λαθρεμπόριο χωρίς να υπάρχει ανάγκη να ε, αποδειχθεί οικονομικό όφελος από αυτή την ε, προσπάθεια. Αντιθέτως, στο πρωτόκολλο των Ηνωμένων Εθνών για το αντίστοιχο θέμα, στο άρθρο 6, αναφέρεται ότι χρειάζεται να υπάρχει οικονομικό όφελος ή κάποιου άλλου είδους υλικό όφελος για να χαρακτηριστεί κάποιος λαθρέμπορος. Παρ' όλα αυτά, στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάποια κράτη-μέλη αποφάσισαν να το δουν διαφορετικά Ακόμα και όταν δεν υπάρχουν ε, κέρδη, ε, έχουν ποινικοποιήσει αυτά τα, αυτές τις πράξεις ε, παρόλο ότι ε, εφαρμόζουν κατά τα άλλα τα, τις του ΟΗΕ. Οπότε τέσσερα μονοκράτη... Γερμανία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο και Πορτογαλία, τηρούν πλήρως τα, τις προδιαγραφές του ΟΗΕ. Μετά υπάρχει άλλο ένα άρθρο που προσδιορίζει τι είναι ποινικό αδίκημα σε ό,τι αφορά την διαμονή ή την παραμονή αλλοδαπών. Ε, εδώ απαιτείται οικονομικό όφελος προκειμένου να χαρακτηριστεί το αδίκημα, ε, η πράξη αυτή ποινικό αδίκημα. Το παράδοξο είναι ότι ε, όταν κάποιοι μετανάστες που ε, ήταν σε τράνζιτ γίνονται μόνιμοι, εκεί μπερδεύονται τα πράγματα. Γιατί Παρόλο ότι απαιτείται οικονομικό όφελος, βλέπουμε ότι 13 από τα 28 κράτη-μέλη θεωρούν, το θεωρούν ποινικό αδίκημα ακόμα και όταν δεν υπάρχει οικονομικό ή υλικό όφελος. Μιλώ για την υποβοήθηση της μόνιμης διαμονής ή παραμονής. Το τελευταίο και πιο σημαντικό άρθρο αφορά το κατά πόσον οι ανθρωπιστικές πράξεις εξαιρούνται. Στο πακέτο της υποβοήθησης λέγεται ότι το κάθε κράτος μέλος θα αποφασίσει αν η ανθρωπιστική συνδρομή θα εξαιρεθεί ή όχι της ποινικοποίησης. Αυτό και αυτό δεν, είναι σε, δεν συμμορφώνεται με τις κατευθείας γραμμές ε, του, των Ηνωμένων Εθνών. Εκεί αναφέρεται το πρωτόκολλο δεν θα απαιτήσει από τα κράτη-μέλη να ποινικοποιήσουν τις πράξεις ομάδων που μεταφέρουν μετανάστες για ανθρωπιστικούς, φιλανθρωπικούς ή αλτρουιστικούς λόγους. Γι' αυτό το λόγο ο ΙΕ πάντοτε επιμένει στην ύπαρξη υλικού ή οικονομικού ωφέλους για να χαρακτηριστεί το αδίκημα λαθρεμπορία προ ή ανθρώπων. Στην, ε, κάποιες ε, ρητές εξαιρέσεις υπάρχουν στις του Βελγίου, της Ελλάδας, της Μάλτας κλπ. Παρ' όλα αυτά, σε αυτές τις εξαιρέσεις, πρώτον, αυτή η εξαίρεση δεν είναι πρώτον ε, υποχρεωτική, δεύτερον δεν εξαιρεί την ανθρωπιστική βοήθεια σε περιπτώσεις ε, διαμονής, τρίτον είναι πολύ περιορισμένες αυτές οι εξαιρέσεις, ε, κυρίως περιορίζεται σε περιπτώσεις ζωής ή θανάτου, επιβίωσης δηλαδή, και ιδιαίτερος ε, όταν προβλέπεται η κατάσταση από το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Δηλαδή κάποιος, κάποιο ε, σκάφος ε, το οποίο βυθίζεται και εκεί χρειάζεται ανθρωπιστικά να διασωθούν ζωές από τον πνιγμό. Τέλος, παρόλο ότι σε ορισμένες χώρες υπάρχουν επίσημες εξαιρέσεις, πολύ συχνά άνθρωποι που προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια ε, κατηγορούνται. Οπότε πρέπει να δει κανένα και το πώ εφαρμόζονται αυτέ οι εξαιρέσει στην πράξη. Αν δούμε τι γίνεται σε όλη την Ευρώπη και θα σας πει περισσότερο συναδελφός μου, ε, άλλο ένα θέμα ήταν το εξής. Δεν είναι σαφές στην Ευρωπαϊκή Ένωση ποιος είναι ο, ο ορισμός της ανθρωπιστικής βοήθειας. Παρ' όλα αυτά, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πάρα πολύ σαφή ορισμό τι είναι ανθρωπιστική βοήθεια στη σχέση τη με τρίτε χώρε. Και το υψηλό επίπεδο κονσένσου τη Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρει ότι η ανθρωπιστική βοήθεια ε, έχει ω ε, στόχο να προσφέρει βοήθεια σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, διατήρηση ε, ε, ε, της ζωής, διατήρηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και όταν οι, τοπικοί, οι τοπικές αρχές δεν μπορούν να ανταποκριθούν επαρκώς. Αυτή η, αυτός ο ορισμός καλύπτει τις περιπτώσεις κρίσης ή τις έκτακτες καταστάσεις στην Ελλάδα και την Ιταλία, για παράδειγμα. Θα μπορούσαμε ενδεχομένω να εμπνευστούμε από αυτόν τον ορισμό. Δεύτερον, θα πρέπει να εμπνευστούμε από την δήλωση ε, του ΟΗΕ για τους, ε, ε, για τα ανθρώπινα, για τους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εκεί λέει ότι οι πολίτες μπορούν να αντιδράσουν στις κρατικές πολιτικές με ειρηνικά μέσα, ιδιαίτερα όταν δρούν προκειμένου να προσπίσουν τα δικαιώματα άλλων. Με άλλα λόγια, όταν οι ακτιβιστές προσπαθούν να υπερασπίσουν δικαιώματα τα οποία καταπατώνται, αυτοί δεν θα πρέπει να, καταδι... διώκονται, αντιθέτως θα πρέπει να θεωρούνται ως υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ακόμα και αν μερικές φορές η δράση τους έρχεται σε αντίθεση με τους κανόνες της, πολιτικής, της μεταναστευτικής πολιτικής ή άλλων πολιτικών σε εθνικό επίπεδο. Οπότε, μήπως θα χρειαστεί κάποια στιγμή να δώσουμε βραβείο Ζαχάροφ σε πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύντομα, που προσπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα πολιτών στην Ευρωπαϊκή, αλλοδαπών πολιτών ενδεχομένω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει λοιπόν να δούμε λίγο και το τι σημαίνει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε Λίνα. Λοιπόν, ο λόγος για τον οποίο επικαιροποιήσαμε την προηγούμενη μελέτη ήταν εν μέρη λόγω της ε, του ταχαιω ρυθμου ρυθμού εξελίξεων 15-16 όταν ολοκληρώσαμε την πρώτη μελέτη. Δηλαδή από τότε μέχρι τώρα και καθότι η πρόσφατη αξιολόγηση κομισιών... είχε λάβει υπόψη τη την προηγούμενη μελέτη μας προσπαθώντα να δει τι άλλο θα μπορούσε να αποσαφηνίσει σε σχέση με την ποινικοποίηση ανθρωπιστικής βοήθειας που έχει σχέση με τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα των πολιτών και την διάσωση της ζωής ε, μεταναστών και προσφύγων. Αναφέρθηκε η συνάδελφος σε κάποιες από τις τυχές αυτές, όπως και στην ε, έλλειψη ασφαλές δικαίου, στις ετερογενείς διατάξεις μεταξύ των κρατών μελών, ως προς κυρώσεις κτλ. Ε, με απογοήτευση σημειώσαμε ότι η αξιολόγηση REFIT δεν φάνηκε να λαμβάνει υπόψη τη πολλές από τις ενδείξεις που εμείς αποστήλαμε, όπως και ακαδημαϊκοί φορείς και οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών προηγουμένω. σχετικά με το γεγονό ότι αυτά τα στοιχεία είναι γνωστά, ευρέω γνωστά και καλά αποδεδειγμένα. Τώρα, είχαμε κάποιες ε, σημαντικές, σοβαρές εξελίξεις σχετικά με την επιβάρυνση της κατάστασης ε, για την ε, ποινικοποίηση ή και την εγκληματική δράση οποιονδήποτε ομάδων ή στο πλαίσιο αυτό θα έχετε ακούσει ίσως τον Καρμέλε Τζούκερο από την Ιταλία τον εισαγγελέα ε, με διάφορες έρευνες που έχουν οδηγηθεί τελικά στην επιβολή ποινικών κυρώσεων σχετικά με ομάδες ε, μη καπαόμικρων εθελοντικές οργανώσεις και τα λοιπά βοηθούσαν για τη διάσωση της ζωής ε, προσφύγων και μεταναστών στην θάλασσα. Η CI, γερμανική μη καπαόμικρον, Τη κατασχέθηκαν τα σκάφη από τη Λιβική εκτοφυλακή. Λιβική εκτοφυλακή που λέγει η ομιλήτρια δεν δρούσε σε, σε συντονισμό με τις επιθυμίες των κρατών μελών που χρηματοδοτούν την επιχείρηση. Και η Κομισιόν μας είπε τελικά Κοιτάξτε, δεν έχουμε τους πόρους που χρειάζεται ή τα μεγέθη που χρειάζονται ε, ώστε να μας δείχνουν ότι ε, ε κλειδώνονται στις φυλακές ε, χιλιάδες χιλιάδων άνθρωποι σε ένα, στα πλαίσια ενός μαζικού φαινομένου διωχμού δηλαδή αν θέλετε να το πούμε έτσι αλλά υπάρχει αντίκτυπος όταν στρέφονται αυτές οι διώξεις κατά των ανθρωπιστικών οργανώσεων. Π.χ. ο Σαλάμ Αλαντίν, με τον οποίο είχα την τιμή να μοιραστώ μια πλατφόρμα, αυτό συνελήφθη στα πλαίσια της δικής του επιχείρησης έρευνας και διάσωσης, φυλακίστηκε και του απαγορεύθηκε η έξοδος από το ελληνικό έδαφος, όπου και συνελήφθη, για ένα χρόνο. Εδώ είναι παράδειγμα ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων τα οποία περιορίζονται και αν θα έλεγα δικαστικής παρενόχλησης παρότι πολλές φορές δεν ολοκληρώνεται η κάθε αυτή νομική αγωγή. Βλέπουμε λοιπόν μία τρομοκρατία που ασκείται και έναν έμεσο διωγμό και παρενόχληση που ασκείται σε οργανώσεις αυτές. Και δεν μιλούμε απλά για διασώστες στη θάλασσα, παρότι είναι από τις πιο σημαντικές θεματικές και πιο συχνές θεματικές. Γνωρίζουμε ότι η Μεσόγειος είναι η πιο επικίνδυνη διέλευση στον κόσμο, αλλά μιλούμε για την παρενόχληση, την ποινικοποίηση διάφορων φορέων ακόμα και σε λίγα χιλιόμετρα από εδώ, στις Βρυξέλλες, όπου καταστρέφονται προσωρινά στρατόπεδα με ε, ε, sleeping bags που έχουν προσφέρει εθελοντές, για παράδειγμα. Και με τις δυνατότητε που δίνονται στις αρχές να προχωρούν σε ε, έρευνες ε, στο χώρο που κατοικούν άνθρωποι εφόσον υπάρχουν υποψίες ότι υπάρχουν εγκληματικά ε, τρομοκρατικές ε, οργανώσεις ή ύποπτοι τέλο πάντων εγκληματικών ενεργειών. Πάρα πολλοί άνθρωποι εκφράζουν μέσω του διαδικτύου την, την επιθυμία τους εθελοντικά να βοηθήσουν πολλούς από τους ανθρώπους αυτούς τους μετανάστες δηλαδή. Επομένως είναι αρκετά σαφέ σε ποιο βαθμό εστιάζεται αυτού του είδους η νομική παρενόχληση αλλά και φορολογική παρενόχληση. Και για να αναφερθώ στην Ουγγαρία βλέπουμε ότι αυτό το πράγμα έχει επιδεινωθεί. Το 2013 όπου ήρθε η κυβέρνηση Φίντες ήδη κυριαρχούσε μια καχυποψία για τις ΜΚΟ που υποτίθεται ότι ήταν ε, τροϊκή ύπη για την εισαγωγή περίεργων ξένων κεφαλαίων τα οποία θα παρενοχλούσαν, θα παρενέβαιναν τέλος πάντων στην εθνική κυριαρχία της χώρας αυξημένες επινές κράτησης για τη διευκόλυνση των δράσεων τέτοιων μη καπαόμικρων, άρνηση χρηματοδότησης και νέα κλιμάκωση του 2018 φέτος για μη κάπα ομικρών που λαμβάνουν εξένη χρηματοδότηση επί της οποίας πρέπει να καταβάλουν πλέον 25% φορολόγηση. Και όσοι λαμβάνουν από ευρωπαϊκούς φορείς ε, στήριξης ε, πρέπει να παραδίδουν τον πλήρη έλεγχο σε κυβερνητικούς φορείς πλέον να αναφερθώ στο σκάφος Aquarius που είναι το μόνο που έχει απομείνει ή στη Μεσόγειο που ενεργεί τέτοιες επιχειρήσεις και ακόμα και σήμερα και χθε αντιμετωπίζει κατηγορίες τύπου ότι ρίχνει απορρίμματα στη θάλασσα κτλ. Δεν είναι μόνο θέμα ελεύθερου είναι και θέμα παρενόχλησης της ίδιας της λειτουργίας καθημερινής των ομάδων των εθελοντικών. Και στην περίπτωση της Ιταλίας ε, χρησιμοποιούνται και διατάξεις ε, νομοθετικές που είχαν εισαχθεί για την καταπολέμηση της μαφίας. Μία από τις συνέπειες είναι ότι τη στιγμή που η Κομισιόν ε, χαίρεται και ικανοποιείται να μειώνει ότι έχουν κατέληθει οι αριθμοί των θανάτων, των μεταναστών, των προσφύγων, θαύμα, αλλά ξέρουμε ότι ο κίνδυνος είναι πιο αυξημένος τώρα. 1 προς 18 είναι αυτή τη στιγμή οι πιθανότητες στη διέλευση της Μεσογείου. Μαζί με τα υπόλοιπα επεισόδια, κρούσματα, κράτησης, απαγωγής, ε, σκαφών των μη καπαομικρών κτλ. Αυτό έχει κινητοποιήσει σε απερίγραπτη κλίμακα τους πολίτες σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Αυτές είναι μόνο κάποιες από τις οργανώσεις που υποστηρίζουν με τη δράση τους. Θα σας παρουσιάσουμε σύντομα και μία, μία, μία ομαδική αναφορά που θα υποβληθεί, που ετοιμάζεται, γιατί είναι θέμα δικαιωμάτων των πολιτών δεν είναι μόνο θέμα μεταναστών ή προσφύγων, είναι θέμα των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών να δρουν σε πνεύμα αλληλεγγύης το οποίο εγγράφεται στις συνθήκες ε, ίδρυσης της Ένωσης. Λοιπόν, αν είναι να αποφύγουμε κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος ε, σχετικά με διώξεις που δεν έχουν κανένα αντικείμενο, και με έναν ευρύτερο κίνδυνο, γιατί νωρίτερα ε, συζητούσατε για, την, ε, για το πόσο υποσκάπτεται η εμπιστοσύνη των πολιτών προ τα θεσμικά όργανα. Είναι θέμα αξιοπιστία και εμπιστοσύνη λοιπόν των ε, θεσμών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα δώσω τώρα λόγο στη Λίνα για κάποιε σύντομε συστάσει. Yeah. So, first... Πρώτη σύσταση λοιπόν, τι δεν πρέπει να ποινικοποιείται. Βλέπουμε πως Πρέπει να εξερεχθούν ε, όσοι έχουν ανθρωπιστική δράση. Σύμφωνα με την οδηγία για την ε, διακίνηση, εξαιρούνται τα θύματα ε, της διακίνησης από την ποινικοποίηση. Οι πρόσφυγες, μετανάστες, διότι στη μελέτη παρέχουμε στοιχεία περιπτώσεων ποινικοποίηση διώξεων και μάλιστα πολλές από αυτές τις περιπτώσεις έχουν οδηγήσει σε καταδίκες. Έπειτα, χρειάζεται έλεγχος, παρακολούθηση της, εφαρμογή, ε, εφαρμογής, διότι βλέπουμε, όπως ακούσαμε και όλες από την Ευρωπαία Λαβήτρια, πως ε, θα μπορούσε, για παράδειγμα, να αναλάβει τον έλεγχο και της παρακολούθησης εφαρμογής των ε, δράσεων περιπτώσεις καταπολέμησης ε, της ε, διακίνησης ανθρώπων, να δούμε τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί, αν έχουμε καταφέρει να ε, διαλύσουμε αυτές τις εγκληματικές οργανώσεις, να τις εξαρθρώσουμε, να δούμε τι μπορεί να γίνει. τι έχουν καταφέρει οι διάφοροι φορείς, όπως για παράδειγμα το Κέντρο Καταπολέμησης της Διακίνησης ε, Ανθρώπων. Επίσης, θα μπορούσε να γίνεται έλεγχος ε, τη συνεργασία ανάμεσα στους ε, διάφορους φορείς, στην κοινωνία των πολιτών, θα μπορούσε να γίνει έλεγχος ε, του αν εφαρμόζονται οι διατάξεις ε, στους ε, συνοριαλικού ελέγχους και επίσης οι αρχές επιβολής του νόμου θα μπορούσαμε να το ζητήσουμε να απαντήσουν σχετικά με το πώς εφαρμόζουν τις οδηγίες και την νομοθεσία. Επίσης υπάρχουν εκρεμείς περιπτώσεις ποινικοποίηση. Υπάρχουν ορισμένες με έντονα πολιτικό χαρακτήρα όπως αυτή που ανέφερε η Τζένιφερ. Σε αυτήν την περίπτωση ίσως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε να, να δημιουργήσει κάποια ε, εξεταστική επιτροπή να δει αν υπάρχουν στοιχεία όπως για παράδειγμα στην περίπτωση του σκάφους Aquarius και εάν οι κατηγορίες που έχουν απαγγελθεί σταθούν. Τρίτη σύσταση. Μακροπρόθεσμη, ολιστική προσέγγιση σε θέματα μετανάστευσης. Πρέπει να ανοίξει πάλι η συζήτηση για την ανθρωπιστική βίζα, ανθρωπιστική θεώρηση. Έχει προταθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η δημιουργία ασφαλών διάβλων εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, επίσης, ε, επιχειρήσεις αναζήτησης και διάσωσης, συνεργασία με την ακτοφυλακή των ε, κρατών μελών. Το λιμενικό σώμα είναι πολύ ε, καλά εξοπλισμένο και ικανότατο για να διεξάγει τέτοιε υπηρεσίες ε, αναζήτηση και διάσωση, έτσι ώστε να σταματήσουν να χάνονται ζωές στη θάλασσα. Προτείνουμε λοιπόν όσοι άνθρωποι διασώζονται από αυτές τις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μετεγκαθίστανται υποχρεωτικά. Αυτά προς το παρόν, τα υπόλοιπα μπορείτε να τα διαβάσετε στην έκθεσή μας, ε, η οποία είναι γεμάτη από στοιχεία. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρωτού δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ήθελα να σκεφτούμε λίγο το τι εστί ε, ανθρωπιά και ανθρωπιστικές αξίες. Νομίζω πως οι λέξεις αυτές έχουν χάσει την αρχική του σημασία και πως ε, είναι πραγματικά τρομακτική η κατάσταση. Το σίγουρο είναι ότι τα παιδιά και τα εγγόνια μας θα κατηγορήσουν εμάς και ως ε, μεμονωμένα άτομα και ως θεσμούς και ως ε, κράτη-μέλη και ως ε, μεμονωμένους υπαλλήλους. Θα μας πούν εσύ τι έκανες για να αποτρέψεις αυτό το κακό εμείς φταίμε, όλοι φταίμε και νομίζω πως πραγματικά χρειάζεται εδώ στην Επιτροπή να νιώσουμε πόσο τρομακτικό είναι αυτό. Πραγματικά αισθάνομαι ντροπή ε, για αυτά που γίνονται στην επικράτειά μας και διάβαζα τώρα πριν από λίγο τι έγινε στην Ιταλία χθες και είναι τρομακτικό, είναι σοκαριστικό. Οι γιατροί χωρίς σύνορα σώζουν ανθρώπινες ζωές στη θάλασσα ε, παίζουν τη ζωή τους κορώνα γράμματα και τώρα μετά ο Σαλβίνη λέει ότι είμαι ε, περήφανος διότι τώρα έκλεισα τα λιμάνια. έχουν γίνει μια σειρά επιθέσεων οι οποίες έχουν στόχο να ποινικοποιήσουν τις ε, επιχειρήσεις διάσωσης ε, στη θάλασσα. Έχουμε χάσει την ανθρωπιά μας και ε, το εννοώ αυτό και το λέω με όλη τη σοβαρότητα. Γι' αυτό λοιπόν τώρα θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μας εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη και πώς φτάσαμε εδώ. Thank you, Mrs. Καταρχήν να ευχαριστήσω τις δύο ερευνήτριε για αυτή την πολύ περιεκτική παρουσίαση. Δεν θα σχολιάσω το περιεχόμενο, διότι μόλις σήμερα το λάβαμε. Να σας πω κάποιες πρώτες παρατηρήσεις όμως. Πρώτη και προφανής παρατήρηση ότι αυτή η μελέτη είναι πολύ χρήσιμη διότι τροφοδοτεί τον προβληματισμό μας. Το πρόβλημά μας είναι σε μεγάλο βαθμό η έλλειψη δεδομένων για την αναμόρφωση του αυτού που ονομάζουμε πακέτο υποβοήθησης. Θα συμφωνήσω σε κάποια πράγματα της μελέτης οπωσδήποτε. Το πρώτο για το οποίο μίλησε και η Πρόεδρος, ότι χρειάζεται αποσαφήνιση των ενιών. Τι είναι λαθρεμπόριο, τι είναι ανθρωπιστική βοήθεια κλπ. Και νομίζω ότι η επικαιροποίηση της μελέτης θα μας διευκρινίσει κάποια πράγματα και αυτό το χρειαζόμαστε. Επίσης, αναφέρατε ότι σε ορισμένες χώρες υφίσταται ακόμα το πρόβλημα της ρήτρα των, της ανθρωπιστικής ακόμα και σε κράτη τα οποία δέχονται εξαίρεση της ανθρωπιστικής βοήθειας από την ποινικοποίηση μερικές φορές ακόμα και εκεί διώκονται τέτοιου είδου ενέργειες. Θα πρέπει να πάρουμε μέτρα έτσι ώστε να αποφεύγουμε τέτοιου είδους διώξεις. Το θέμα της ανθρωπιστικής βοήθειας επίσης δεν έχει να κάνει μόνο με τη θάλασσα. Ε, μιλάμε πολύ για τη θάλασσα γιατί τέτοιου είδους επεισόδια βλέπουμε πολύ συχνά στα μέσα ε, ενημέρωσης. Ε, αλλά η ανθρωπιστική βοήθεια δίδεται σε διάφορες άλλες και σε διάφορες άλλες περιπτώσεις. Επίσης πρέπει να δούμε τι συμβαίνει σήμερα. Βλέπουμε διάφορες μαρτυρίες στα μέσα ενημέρωσης. Όπως έχουμε καταλάβει, χρησιμοποιούνται και άλλοι νόμοι, άλλου τύπου νομοθεσία για να διωχθούν ανθρωπιστικές οργανώσεις. Όπως είδαμε για παράδειγμα, χρησιμοποιήθηκε ένας νόμος κατά της μόλυσης της θάλασσας πρόσφατα. Πρέπει ενδεχομένω να δούμε και τις άλλες πτυχές της νομοθεσίας λοιπόν. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Για όσους δεν θυμόμαστε να σας θυμίσω ότι εμείς ζητήσαμε την αρχική μελέτη το 2016. Μετά η Κομισιόν έκανε μια αξιολόγηση refit όλης οδηγίας, αλλά αποφάσισε προς το παρόν να μην την τροποποιήσει. Η ερώτηση είναι γιατί. Γιατί να μην εξασφαλίσουμε νομική ασφάλεια. στην οδηγία. Και ακόμα δεν μας έχει απαντήσει η Κομισιόν σε αυτό το ερώτημα. Οπότε ζητήσαμε από το ε, Policy Department ε, C του Κοινοβουλίου να επικαιροποιηθεί αυτή η μελέτη. Και τώρα, σύμφωνα με τα πορίσματα, θα πρέπει να προσαρμοστεί, να τροποποιηθεί και η οδηγία για την υποβοήθηση. Πολλοί από εμάς μεταξύ και αυτών και εγώ ίδια, θα είχαμε καταδικαστεί στο παρελθόν για βοήθεια που έχουμε δώσει σε ανθρώπους. Πολλά χρόνια πριν βέβαια, δεν χρειάζεται να κάνεις να φωνάξει στην αστυνομία, έχουν παραγραφεί αυτά τα δικήματα. Αυτό που λέω όμως είναι ότι έχουμε, είμαστε ακόμα άνθρωποι ή έχουμε γίνει ρομπότ. Καλή ερώτηση. I have to leave. in 10 minutes. Πρέπει να ε, σας πω ότι θα έχουμε και μια ομάδα επισκεπτών σε λίγο. Να πω καταρχάς ότι ε, θέλω να ευχαριστήσω τη Σεσίλια για το ότι ήσουν σαφέστα, σαφέστατη. Και μάλιστα στα Δανέζικα είναι ακόμα ε, πιο ενδιαφέροντα αυτά που είπες ε, λόγω της ε, μικρής διαφοράς της γλώσσας. Πραγματικά ποιος μπορεί να βλέπει αυτά που γίνονται και να μένει απαθής. Ε, πρέπει να είναι άκαρδος κάποιος για να μην συγκινηθεί, για να μην σοκαριστεί. Φυσικά έχουμε κάποιες αξίες τις οποίες πρέπει να τηρούμε. Δεν είναι δυνατόν όταν υπάρχει το δίκαιο της ε, θάλασσας ε, να μιλάμε για τέτοια πράγματα. Θυμάμαι πως όλα τα σκάφη όταν συναντούσαν έναν ναυαγό, έναν άνθρωπο στη θάλασσα, ήταν καθήκον τους να τον διασώσουν και αυτό το έμαθα παιδί ακόμα. Και μάλιστα ως ε, Δανέζα έχουμε εμπειρία στη διάσωση. Είχαν διασωθεί πάρα πολλοί Εβραίοι και πέρασαν από τη Δανία στην Σουηδία ήταν μια πανάκριβη επιχείρηση διάσωσης ε, και δεν το λέω για το οικονομικό κόστος, αλλά η όλη η επιχείρηση του να, τους, να βάλουν αυτούς τους ανθρώπους ε, στις ε, βάρκες, στα σκάφη και να τους περάσουν απέναντι στη Σουηδία είχε κοστίσει. Φανταστείτε τι θα μας έλεγαν, αν αυτό γινόταν τώρα, το 2018, θα μας έλεγαν ότι διακινούμε ανθρώπους. Θα μας θεωρούσαν εγκληματίες. Πολύ σωστά τα είπες, Σεσίλια. Δεν πρέπει να κατηγορούμε τους ε, Ιταλούς. Όμως πρέπει να παραδεχτούμε ότι υπάρχει έλλειψη αλληλεγγύης στην Ευρώπη και νομίζω ότι στην έκθεσή σου προς ε, ε, το Συμβουλίο αναφέρθηκες με πολύ σωστά λόγια. Η αλληλεγγύη πρέπει να προέρχεται από όλα τα κράτη-μέλη. Όλοι πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους ε, και το μερίδιο που τους ε, αναλογεί. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τι συμβαίνει. Νομίζω πως πρέπει να συνεχίσουμε να μιλάμε με λόγια στα ράτα και να προφυλάσσουμε τις ε, αξίες, την ανθρωπιά μας, διότι η ανθρώπινη ζωή είναι αυτό που μετράει πάνω από οτιδήποτε άλλο. Ευχαριστώ πολύ Μάργαρετ, σας ευχαριστώ πολύ όλους. Ε, θα επανέλθουμε, σας το υπόσχομαι, πολύ σύντομα ε, στο θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν. Νομίζω πως ε, τώρα έχει έρθει η ώρα να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης. Ας πάρουμε όμως μία ανάσα γιατί νιώθω πραγματικά πως είμαι σε κατάσταση σοκ. Έχω αδειάσει από όλα αυτά που άκουσα. Υπάρχουν... Γίνεται ένας αγώνας προς τον πάτο πραγματικά και ελπίζω αυτό να μην γενικευθεί και στα θεσμικά όργανα. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημέρας διάταξης, ε, το σημείο 18, αναφορά 1247, στο ίδιο θέμα. Είναι μαζί μας η αναφέρουσα Πάουλα Σμιτ Πόρας σας καλωσορίζω στην Επιτροπή και σας δίνω το λόγο για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Βίξτρομ, ευχαριστώ πολύ που με δέχεστε πάλι στην Επιτροπή σας. Και ευχαριστώ πολύ την Επιτροπή Αναφορών που ασχολείται με την ε, αναφορά μου για δεύτερη φορά. Δεν είμαι εδώ για την περίπτωση των τριών πυροσβεστών που, δόξα τω Θεώ, αθώθηκαν. Θέλω να σας επιστήσω την προσοχή στην περίπτωση του Σον Πάιντερ και της Σάρα Μαρντίνη, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι στην Ελλάδα σε μια φυλακή ε, υψηλή ασφάλεια και κατηγορούνται για το ίδιο πράγμα, για ε, εμπορία ανθρώπων, για διακίνηση ανθρώπων ένας από αυτούς είναι, ε, είναι πρέσβυρα καλής θέλησης στα Ηνωμένα Έθνη και αυτές οι κατηγορίες ολοένα ε, και σοβαρεύουν, γίνονται ένα και πιο βαριές. Γι' αυτό λοιπόν θα περάσω κατευθείαν στην παρουσίασή μου, την οποία έχω προετοιμάσει για να με βοηθήσει. Και ελπίζω αυτό να μην προσμετράτε στα πέντε λεπτά που έχω για να παρουσιάσω την αναφορά. Έχουν μείνει τέσσερα λεπτά. Γι' αυτό λοιπόν ζητώ συγγνώμη από τους διερμηνείς επειδή θα μιλήσω πάρα πολύ γρήγορα. Now, are we the committee fit for purpose this afternoon? <laughs> Δεν ξέρω αν η Επιτροπή μας μπορεί να ταπεξέλθει στις προσδοκίες ε, σας σήμερα το απόγευμα. Νομίζετε πως δεν είναι καλό να αρχίσετε. Ναι, ναι, αλλά θέλω να αρχίσω, αλλά νομίζω πως ε, θα βοηθήσει αν έχουμε και οπτικό υλικό. Ναι, λέει πρόεδρο, αλλά πόσο χρόνο χρειάζονται οι τεχνικοί για να στήσουν την παρουσίαση. Meanwhile, could you give me... Ωραία, θα μπορούσατε να μου πείτε ξανά το όνομα της ε, Σάρα. Ναι, Σάρα Μαρντίνη είναι πρόσφυγας από τη Συρία η οποία έγινε γνωστή πριν από δύο χρόνια διότι κολύμπησε με την αδελφή της από την Τουρκία στην Ελλάδα. Ε, ήταν πάνω σε, μια βάρκα με άλλους ε, Σύρους πρόσφυγες. Η βάρκα καταστράφηκε και 17 άτομα πάνω στη βάρκα ε, πέσαν στη θάλασσα που δεν είχα, που, και δεν ήξεραν κολύμπη και μια που η Σοφία και η αδελφή της ήταν επαγγελματίες, κολυμβήτριες, κολύμπησαν για 7-8 ώρες συνεχόμενες και έσπροχναν την ε, βάρκα ε, που είχε καταστραφεί προς τις ελληνικές ακτές. Όπως σας είπα, έγιναν διάσημες. Η μία έγινε πρέσβυρα καλής θέλησης στην ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Πήγαν και οι δύο στους, στους Ολυμπιακούς Αγώνες με την ομάδα των προσφύγων. Και συμμετέχουν ενεργά στη, στα θέματα της ανθρωπιστικής κρίσης ε, στην Ελλάδα και τώρα εκρεμούν κατηγορίες που εφόσον ε, καταδικαστούν ε, θα φυλακιστούν για 15 χρόνια. Οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Υπάρχουν επίσης 7 ε, εργαζόμενοι στον ανθρωπιστικό τομέα οι οποίοι εμπλέκονται στις ε, κατηγορίες αυτές η κατάσταση ολοένα και χειροτερεύει για τους ε, επαγγελματίες, για τους εργαζόμενους ανθρωπιστικές οργανώσεις και για όσους βοηθούν μετανάστες νόμιμους ή μη για ανθρωπιστικούς λόγους. Δεν έχει καμία σημασία το πώς εισέρχεται κάποιος στη χώρα. Η βοήθεια έχει ανθρωπιστικούς λόγους. Οι κατηγορίες λοιπόν που τους βαρύνουν ολοένα και επιδεινώνονται. Όπως σας είπα είναι προφυλακισμένοι και περιμένουν τη δίκη τους. Μπορείτε να μας γράψετε τα ονόματα. Ναι, Σάρα Μαρντίνη και να μας πείτε σε ποια φυλακή βρίσκονται όλες οι σχετικές λεπτομέρειες και να μου δώσετε αυτές τις πληροφορίες. Είμαστε έτοιμοι τώρα. Ναι, Σάρα Μαρντίνη και Σον Μπάιντερ ονομάζονται. Δεν είναι οι μόνοι όμως. Θα ήθελα να μάθω σε ποια φυλακή κρατούνται και μπορεί να μεταβούμε εκεί αν γίνεται. Μπορώ να πάω και μόνη μου. Ναι, πέντε διαφάνειες έχω να σας δείξω μόνο γιατί έχω πέντε λεπτά. Νομίζω πως θα σας βοηθήσουν όμως ε, να καταλάβετε το τι συμβαίνει στις αίθουσες των δικαστηρίων. Μάλλον υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα και δεν γίνεται να δείξουμε τις διαφάνειές σας. Γι' αυτό λοιπόν ε, θα αναγκαστείτε να μιλήσετε χωρίς αυτές. Σίγουρα μπορείτε και έχετε ε, την κατάλληλη εφράδια για να το κάνετε. Θα προτιμούσα να περιμένω αν έχουμε την ελπίδα θα φτιαχτεί, αλλά δεν έχουμε χρόνο, λέει η πρόεδρο. Οπότε θα είναι λίγο πιο περίπλοκη η παρουσίασή μου. Θα, μπορώ, θα μπορούσα να σας στείλω με email την ε, παρουσίασή μου. Δεν την έχω καν μπροστά μου, της διαφάνειες εννοώ. Το βασικό όμως θέμα είναι ότι τα δύο τελευταία χρόνια πολλά έχουν γίνει. Η κατάσταση είχε εξελιχθεί. Η αξιολόγηση refit της Κομισιόν είναι πολύ απογοητευτική. Όχι, δεν είναι αυτή η παρουσίασή μου. Αυτή είναι η παλιά μου. Αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Ε, χαίρομαι που, τα, έχουν, την έχουν ευρωβουλευτές τουλάχιστον. Ε, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, δηλαδή δικηγόροι, ε, υπεράσπισης, οι ερευνητές, οι, ε, οι ακτιβιστές κλπ. Ακόμα η ΟΚΕΟΙΕ το 18, η Κομισιόν, όλοι οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να αλλάχθει να αλλάξει το άρθρο 1 παράγραφος 2 του πακέτου υποβοήθησης. Γιατί, γιατί πολύ απλά πρόκειται για παραβίαση του Ευρωπαϊκού Χάρτη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου. Α, ωραία, τέλεια. Εδώ είναι η παρουσίασή μου. Αυτή είναι η, μία από τις αδελφές της Σάρα, τη Σάρα Μαρντίνη, που ζητάει την απελευθέρωσή της. Έλεγα λοιπόν ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς συστούν την τροποποίηση του άρθρου 1 παράφως 2. Η αξιολόγηση refit είναι πάρα πολύ απογοητευτική, γιατί δεν εντόπισαν δεδομένα. Δεν ξέρω πώς κάνουν την έρευνά τους, Λένε ότι δεν υπάρχουν αρκετέ περιπτώσει ποινικοποίηση τη ανθρωπιστικής βοήθειας, Θεωρούν ότι αναγνωρίζουν ότι το πακέτο δεν ήταν αποτελεσματικό ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη διάκριση ανάμεσα στην ανθρωπιστική βοήθεια και, την, και το ποινικό αδίκημα, αλλά δεν θέλουν να το τροποποιήσουν παρόλα αυτά. Και ένα άλλο θέμα, ακόμα και τα 7 κράτη-μέλη τα οποία έχουν μεταγράψει την οδηγία, τους στις εθνικές, την οδηγία ακόμα και αυτέ οι χώρε και σε αυτέ τι χώρε οι εισαγγελείς έχουν βρει τρόπου να ποινικοποιήσουν τι συγκεκριμένε δράσει, Οπότε και πάλι δεν έχουμε ε, εγγύηση για την ασφάλεια των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Όπως είπατε και εσείς, η Κομισιόν αποφάσισε να διατηρήσει την νομοθεσία όπως έχει. Θεωρώ ότι είναι σκανδαλώδε. και η Κομισιόν λέει ότι παρόλο ότι υπάρχουν κίνδυνοι ποινικοποίηση ανθρωπιστικής βοήθειας, δεν θεωρεί ότι αυτοί οι κίνδυνοι σχετίζονται ιδιαίτερα με το νομικό πλαίσιο. Για μένα ως δικηγόρου αυτό είναι σκανδαλώδες διότι έχουμε εντοπίσει πάνω από 80 περιπτώσεις ποινικοποίηση δράσης των ε, πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βοηθούν ε, παράτυπους μετανάστες ή ετούντες ε, διεθνούς προστασίας όλα τα ψηφίσματα, οι κώδικες, οι συναντήσεις με τους εμπλεκόμενους κλπ. Όλα αυτά πολύ καλά και ευχαριστούμε πάρα πολύ και για το ψήφισμα του Αυγούστου 2018, αλλά τίποτα από αυτά δεν είναι δεσμευτικό νομικά. Τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι οι δικαστές δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν όλα αυτά στις δικαστικές διαδικασίες, διότι οι δικαστές εφαρμόζουν μόνο τον νόμο σε συνδυασμό με τα τεκμήρια και τις, α, ε, τα στοιχεία που διαθέτουν. Άρθρο 214 της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης λέει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να καθορίσει το πλαίσιο των ανθρωπιστικών δράσεων και οι ανθρωπιστικές δράσεις θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα με βάση τις αρχές του διεθνούς δικαίου. Αυτό είναι ο δικός σας ρόλος. Γιορτάζουμε τα 70 χρόνια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η συνθήκη τη Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται πάνω στην αρχή τη ανθρώπινη αξιοπρέπεια, του κράτου δικαίου, τη δικαιοσύνη και της αλληλεγγύη. Και τι ζητάμε, ζητάμε να αλλάξει μόνο μία λέξη, το άρθρο 1-2. Εκεί που λέει το κράτο μέλο δύναται να αποφασίσει να μην και λοιπά, να γίνει σαλ αντί για may, δηλαδή το κράτος μέλος αποφασίζει ή δέον να αποφασίσει να μην κλπ. κλπ. Να μην ποινικοποιήσει δηλαδή την ανθρωπιστική βοήθεια. Ευχαριστώ. Ε... Εγώ σας ευχαριστώ λέει Πρόεδρος. Νομίζω ότι με μεγάλο ενδιαφέρον θα ακούσουμε τώρα την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρακαλώ. Έχετε το λόγο ιδιαίτερα, ιδιαίτερα σε αυτό. Τη ρήτρα ΣΕΙ Σαλ ή Μέι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και τους υποβάλλοντες. Ευχαριστούμε για την παρουσίαση αυτή. Χαίρομαι που ακούω ότι οι πελάτες σας κρίθηκαν αθώοι. Ήταν μια έκκληση που απευθύναμε διαρκώς χωρίς ανταπόκριση μέχρι και την προηγούμενη φορά, δηλαδή να μας ενημερώνετε με όλες εκείνες τις περιπτώσεις καταδίκης <clears throat> στις οποίες αναφέρεστε, αυτές τις 80 δηλαδή περιπτώσεις, υποθέσεις. Γιατί είναι κρίσιμη σημασία για εμάς να έχουμε τα στοιχεία, εφόσον μας έχουν διαφύγει, για να τα εξετάσουμε. Σας παρακαλώ λοιπόν να μας δίνετε αυτές τις πληροφορίες, να μας δώσετε αυτές τις πληροφορίες. Από την τελευταία φορά που είχαμε συναντηθεί, η θέση της ε, Επιτροπής δεν έχει μεταβληθεί, δεν θα επαναλάβω δηλαδή <clears throat> αυτά που είχαμε πει. Πέραν του ότι θα πω, ότι θυμίζουμε διαρκώς το γεγονός ότι σε καμία περίπτωση η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία δεν ποινικοποιεί την ανθρωπιστική βοήθεια. Είχαμε τακτικέ επαφέ με όλου τους ενδιαφερόμενου φορείς, γιατί παρά το γεγονό ότι το συμπέρασμα του Refit ήταν ότι δεν χρειάζεται νομοθετική επανεξέταση, έλεγε ότι υπάρχει όχι μόνο απευθεία ο κίνδυνος της ποινικοποίηση, αλλά και η αίσθηση, η εντύπωση του κινδύνου ή και της αγωγής, όχι μόνο της ποινικοποίηση. Όπου και να οδηγεί δηλαδή αυτή. Και στην αξιολόγηση refit είχαμε δεσμευθεί ότι θα συμμετάσχουμε, θα συνεργαστούμε στενά με όλους τους ενδιαφερόμενους για να δούμε πώς θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε το θέμα. Και αυτό κάναμε. Διοργανώσαμε μια συνέντευξη τον περασμένο Μάιο με όλους τους ενδιαφερόμενους και με την ΣΕΠΣ για μια πρώτη επικαιροποίηση και μία από τις προτάσεις ήταν να διατεθεί μια ψηφιακή πλατφόρμα σε όλους τους μη και να ανοίξουμε την διαθεσιμότητα αυτή, δηλαδή να διαθέσουμε μάλλον την δυνατότητα αυτή σε όλους τους μη ομικρών τους ενδιαφερόμενους με μια δυνατότητα τμήματος για τα κράτη-μέλη όπου ο καθένας θα μπορούσε να τροφοδοτεί την πλατφόρμα αυτή με τις πληροφορίες και τις ενδείξεις εκείνες που ακόμα μας λείπουν. Μέχρι στιγμής δεν λάβαμε καμία θετική ανταπόκριση ή απάντηση, αλλά θα επαναλάμβανα την πρόσκλησή μας να το πράξετε αυτό. Συναντηθήκαμε επίσης με τη Eurojust, με μια συνάντηση το Μάιο επίσης ε, μεταξύ ειδικευμένων τμήματων εισαγγελία και ανακριτών που ερευνούν τέτοια θέματα και με τη σκέψη ίσως δημιουργίας μια συγκεκριμένη ε, task force που θα ήταν αφιερωμένη σε αυτή τη δουλειά. Επίσης ακούσαμε ότι η ΦΡΑ, λέει η ομιλήτρια, έχει προχωρήσει σε μια δουλειά όλων των υποθέσεων ποινικοποίηση που αφορούσαν σε επιχειρήσεις ε, έρευνας και διάσωσης στην Μεσαιόγειο θάλασσα. Σας ευχαριστώ λέει ο Για το σαλ email που σας ζήτησα, απάντηση δεν έχουμε. Μάλλον δεν έχουμε, οπότε απλώς θα σημειώσουμε ότι δεν έχουμε. Οπότε τώρα θα δώσω το λόγο στα μέλη. Η κυρία Καβεθόν Ρουίθ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ξεκινούσα ευχαριστώντας τους ε, αναφορείς τους αναφέροντες, με συγχωρείτε. Είχαμε και την περίπτωση των πέντε πυροσβεστών από την Σεβίλη που είχαν θέσει το... που είχαν κάνει την αρχική ε, καταγγελία. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμη η αναφορά αυτή, διότι υπάρχει μια έλλειψη ασφάλειας δικαίου. Η Κομισιόν μας είπε ότι δεν βλέπει πρόβλημα ερμηνείας νομικής, αν όμως δεν υπάρχει πρόβλημα ε, νομικής ερμηνείας, ίσως μας λείπουν μηχανισμοί. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρχει κανένα είδου αποδοχή φαινομένων ποινικοποίηση ανθρωπιστική βοήθεια. Και επομένω, εφόσον δεν υπάρχει δυσκολία, αναστολή νομικής ερμηνεία, θα έπρεπε να έχουν αναπτύξει μηχανισμούς κυρώσεων που δεν έχει γίνει και επομένως κάτι δεν είναι σαφές. Δηλαδή είτε η οδηγία αυτή δεν δημιουργεί την ασφαλεία δικαίου που χρειάζεται ή δεν ερμηνεύεται επαρκώς από τα κράτη-μέλη. Σε οποιαδήποτε από τις δύο περιπτώσεις κάτι πρέπει να γίνει. Και έχω την εντύπωση, λόγω της σοβαρότητας του θέματος, που δυστυχώς δεν απασχολεί, δεν μας απασχολεί τόσο, δεν έρχεται στην επιφάνεια τόσο συχνά στις δικές μας ακτές τουλάχιστον. Θα έπρεπε ίσως από την Επιτροπή των Ελευθεριών και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γενικώ θα έπρεπε να ασκηθεί μια πίεση ή να αναλυθεί κάποιο άλλο μέτρο ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την οδηγία αυτή εφόσον χρειάζεται κάποια βελτίωση προκειμένου να ερμηνεύεται πλήρως και να παρέχει νομική ασφάλεια. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Βαλίνα, η Μπεατρίση επίσης ζήτησε το λόγο. Α, τότε μετά την Άντζελα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήδη από το προηγούμενο σημείο μιλούσαμε για την έλλειψη αξιοπιστία και την ε, όλο και μεγαλύτερη καχυποψία ή έλλειψη έλλειψη εμπιστοσύνη από πλευρά των πολιτών. Και εδώ έχουμε ένα από τα πιο σοβαρά κρούσματα προς την κατεύθυνση αυτή. Ε, κάποιοι αναρωτιούνταν αν έχουμε γίνει ρομπότ, αλλά εδώ μιλούμε όχι για ρομπότ, αλλά για ε, μεταμόρφωση σε εγκληματικά στοιχεία. Δηλαδή αυτό ονομάζεται δολοφονία. Εάν δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο της ποινικοποίησης των ανθρώπων αυτών που προσπαθούν να αποτρίψουν τον χαμό ανθρωπίνων ζώων, ε, τότε πρέπει να μιλούμε για δολοφονία. Δεν πληρούμε τις διεθνείς μας υποχρεώσεις. Δεν ξέρω αν αυτή η οδηγία είναι εδώ για να ακυρώσει διεθνείς συνθήκες για τη θάλασσα. Είμαστε σε απόλυτη αντίφαση προς την Χάρτα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Δηλαδή αντιτίθεται προς τα πάντα. Και μετά διαμαρτυρόμαστε που ε, κερδίζει έδαφος ε, ο φασισμός και τα λοιπά λέει η ομιλήτρια. Οι διεθνείς μας υποχρεώσεις είναι ο σεβασμός της ανθρώπινης ζωής, των πολιτών και των οργανώσεων που δρούν για να σώζουν τις ζωές των ανθρώπων αυτών που έρχονται με τρόπο άτυπο και που ποτέ δεν θα έπρεπε και ποτέ δεν πρέπει να τους θεωρούμε παράνομους όπως πολλοί λένε. Νομίζω ότι χρειάζεται ανάληψη επίγουσα ανάληψη δράσης για την οδηγία αυτή προκειμένου να συμμορφωνόμαστε προς το διεθνές δίκαιο των θεμελιωδών δικαιωμάτων, την διεθνή συνθήκη για το δίκαιο της θάλασσας, τη διεθνή συνθήκη για την καταπολέμηση του λαθρομπορίου ανθρώπων, την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις συνθήκες τις ιδρυτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τις έχουμε ξεχάσει σε ένα σκοτεινό σιρτάρι. Κάθε μέρα που περνάει είναι μια ακόμα χαμένη ημέρα και διάφορες ακόμα χαμένες ζωές ανθρώπινες. Είναι προφανές ότι οι αναφέροντες εντοπίζουν ένα ξεκάθαρα υφιστάμενο πρόβλημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι, φαίνεται αδύναμη να εγγυηθεί οτιδήποτε. Φαίνεται να είμαστε ικανοί να δημιουργήσουμε συγκρούσεις, να στήσουμε συγκρούσεις σε διάφορα μέρη του κόσμου, αλλά όχι να προασπιστούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι πρώην λαθρέμποροι τώρα είναι ακτοφύλακες. Αυτό σκεφτείτε. Και ποιος εμπορεύεται το πετρελαιό τους. Αυτό δεν θέλουμε να το πούμε έτσι, μάλλον όχι. Εγώ ε, θεωρώ ότι αυτή η αναφορά πρέπει να μείνει ανοιχτή. Θεωρώ ότι η Κομισιόν πρέπει να απαντήσει γραπτός, γραπτός και ότι η Επιτροπή μας θα πρέπει να υποβάλει προφορική ερώτηση με ψήφισμα για την Ολομέλεια ώστε να τοποθετηθεί το Κοινοβούλιο προκειμένου η Κομισιόν να προχωρήσει σε τροποποίηση της οδηγίας αυτής άμεσα δεν μπορούμε να επιτρέψουμε το φαινόμενο αυτό να συνεχιστεί. Ευχαριστώ. Thank you very much, Η Άγγελα Βεατρίθ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, λυπάμαι που βλέπω σαν προσώπους της Κομισιόν, γιατί έχουμε άλλο ένα πολύ σοβαρό κρούσμα που μας αποδεικνύει ότι τα πράγματα δεν έχουν επιληθεί ότι δεν έχουμε βρει λύση, όλα αυτά είναι πολύ νεφελώδη για εμάς. Προφανώς και εγώ είμαι κατά της ποινικοποίησης της ανθρωπιστικής βοήθειας και των οργανώσεων, αλλά επίσης είμαι και κατά της ε, ποινικοποίησης εντός των προσπαθειών που μπορεί να καταβάλει και καταβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε κενά τα κενά μας είναι στον συντονισμό και στη συμμόρφωση προς το εθνές δίκαιο. Και τα κενά μας αυτά, οι απώλειες αυτές, σημαίνουν ανθρώπινες ζωές. Έχουμε δράση ανθρωπιστικών οργανώσεων, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, οργανώσεων υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η, περασμένη εβδομάδα ε, ήταν ξεκάθαρη ως αυτό, μας το είπε και η ίδια η καγκελάριος Μέρκελ. Είχαμε την επιχείρηση Τρίτων, την επιχείρηση Σοφία. Ε, φαίνεται ότι τα κράτη-μέλη σε καμία περίπτωση δεν είναι σε θέση να φτάσουν σε μια συμφωνία. Η κυρία Μογκερίνη προσπαθεί να ξεμπλοκάρει την κατάσταση. Ε, οι επιχειρήσει αυτέ ε, έσωσαν 200.000 ανθρώπινε ζωέ στην Μεσόγειο. Αλλά αυτά είναι ανυπαρκή. Και είναι σαφέ. Και υπάρχει και άλλο ένα σαφές σημείο. Αν δεν είμαστε ικανοί να αλλάξουμε εδώ μία λέξη, τι είμαστε ικανοί να κάνουμε. Εδώ μιλάμε για την αντικατάσταση του ΜΕΙ από το ΣΑΛ. Το εθελοντικό που υπάγεται στα μικροκομματικά και άλλα ωφέλη ή συμφέρον με το ΣΑΛ που σημαίνει υποχρέωση. Εγώ νομίζω ότι η αναφορά πρέπει να συνεχίσει. Πρέπει να σας ε, πω πως έχουμε ξεφύγει τελείως από το χρονοδιάγραμμά μας. Πρέπει να συντομεύουμε. Και μια που ξεκινήσαμε πολύ αργά, είμαι σίγουρη, Παόλα, ότι μπορείς να συνοψίσεις μέσα σε ένα λεπτό. Ναι, θα, σας ευχαριστήσω όλους για τη στήριξη που δείχνετε. Και νομίζω ότι όταν προσπαθούμε να αλλάξουμε το κόσμο πολύ συχνά καταφέρνουμε να έχουμε και τον ε, κατάλληλο αντίκτυπο. Προσπαθούμε να αλλάξουμε την νομοθεσία, ωστόσο χρειάζεται ένα νομικό πλαίσιο για την ανθρωπιστική βοήθεια στην Ένωση. Το πλαίσιο αυτό δεν υπάρχει ακόμα, δεν έχει αναπτυχθεί επαρκώς και νομίζω ότι το άρθρο 214 που αναφέρεται στις επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας είναι ελλειπές όλο το βάρος δόθηκε στην ε, πολιτική κατά της ε, διακίνησης του, του λαθρεμπορίου ανθρώπων. Έχω δει με τα μάτια μου θύματα διακίνησης ε, ανθρώπων και άκουσα φρικιαστικές ιστορίες τι τραβάνα μέχρι να φτάσουν στην Ευρώπη. Ωστόσο, οι, επιχει... οι ανθρωπιστικές επιχειρήσεις πρέπει να πλαισιώνονται με σαφήνεια. Πρέπει να υπάρχει προστασία, διεθνής προστασία για εκείνους που ε, την χρειάζονται. Ε, δεν έχει σημασία αν είναι μετανάστες ή πρόσφυγες, έχουν κάποιο λόγο που ε, κάνουν αυτό το ταξίδι, αλλά και να προστατεύονται οι εργαζόμενοι ε, στον ανθρωπιστικό κλάδο και όχι μόνο αυτοί, όλοι οι άνθρωποι που δείχνουν ανθρωπιά και αλληλεγγύη και προσπαθούν να βοηθήσουν ανθρώπους που έχουν ανάγκη και βρίσκονται σε πολύ άσχημη θέση διότι είναι παράτυποι, δεν μπορούν να νοικιάσουν σπίτι, δεν μπορούν να βρουν δουλειά, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Πρέπει να βασιστούμε στις ευρωπαϊκές αξίες τις οποίες μοιραζόμαστε, τις οποίες έχουμε κοινέ ε, στην Ευρώπη. Υπάρχουν πάρα πολλέ περιπτώσεις, όχι μόνο σε μη κυβερνητικέ οργανώσεις, αλλά και μεμονωμένοι πολίτες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή ε, αντιμετωπίζουν βαρύτατε κατηγορίες για ε, το ότι βοήθησαν άλλους ανθρώπους. Σα ευχαριστώ πολύ. Φυσικά θα μείνει ανοιχτή αναφορά και νομίζω πως ε, θα έπρεπε να στείλουμε μια επιστολή στην κυβέρνηση της Ιταλίας, διότι αυτό που έγινε, εκτός από αυτά που διαβάσαμε στις ε, εφημερίδες, είναι σοκαριστικό, είναι απίστευτο. Ναι, και στην ελληνική κυβέρνηση φυσικά. Ναι, και στις ε, ελληνικές αρχές ε, για την περίπτωση Σάρα Μαλτίνη και Σον Μπάιντερ. Να δούμε πού κρατούνται, υπό ποιε συνθήκες και ε, πώς προχωράει η περίπτωσή τους. Ελπίζω να καταφέρουμε να επιτύχουμε κάτι. Ωστόσο, το θέμα μας εδώ είναι ότι πρέπει να στείλουμε μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Δημήτρη Αβραμόπουλο προσωπικά. Ε, πρέπει να λάβει μία επιστολή γραμμένη με ομά ε, λόγια για να ε, θέσουμε την κατάσταση και να ζητήσουμε να υπάρχει αυτή η εξαίρεση για την ανθρωπιστική βοήθεια, δηλαδή ό,τι προβλέπει η οδηγία. Και επίσης να ξεκινήσει πολύ γρήγορα η διαδικασία τροποποίησης της οδηγίας, μια που η τροποποίηση είναι πάρα πολύ μικρή. Όμως, επαναλαμβάνω ότι αυτή η αναφορά είναι μία από τις σημαντικότερες που έχουμε αναλάβει ως Επιτροπή φέτος και ίσως σε όλη τη διάρκεια της θητείας μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν που τονίσατε την ε, σημασία αυτής της αναφοράς και ε, ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να, ε, να ενημερωθεί για το πόσο σημαντικά είναι τα πράγματα. Σας ευχαριστώ πολύ που δραστηριοποιήσετε την ανθρωπιστική βοήθεια και που ήρθατε εδώ να μας παρουσιάσετε το τι συμβαίνει. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους και έχει έρθει η ώρα να περάσουμε στην επόμενη αναφορά. 420 για τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Δεν είναι μια συμφωνία, είναι μια δήλωση εδώ που τα λέμε. Ε, έχει την ίδια νομική βαρύτητα με ένα ανακοινωθέν τύπου. Ο αναφέρον δεν είναι εδώ, όμως έχουμε τον εκπρόσωπο τον κύριο Ράιον, ο οποίος θα λάβει αμέσως το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημοσιεύσει τις παρατηρήσεις της το Μάιο του 2018. Μας ζητήθηκε να παράσχουμε λοιπόν ε, τις παρατηρήσεις μας. Η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας ολοκληρώθηκε το Μάρτιο του 2016 και ε, είναι πλήρως συμμορφούμενη με το ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο. Επιτρέπει την επιστροφή μεταναστών οι οποίοι έχουν εισέλθει παράτυπα ε, αλλά και ε, περιπτώσεις σε τον άσυλο των οποίων οι αιτήσει έχουν απορριφθεί. Αυτή η πτυχή είναι εκείνη στην οποία ασκήθηκε η δρυμύτερη κριτική από τον αναφέροντα. Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι από την ε, πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η ασφάλεια, η κατάσταση ασφαλείας στην Τουρκία πρέπει να ε, εξεταστεί και συνολικά αλλά και μεμονωμένα. Οι αρχές ε, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να είναι σίγουρες ε, μεν ότι η κατάσταση στην Τουρκία είναι ασφαλής αλλά και για τον αναφέροντα να πούμε ότι η συμφωνία προβλέπει ότι η χρήση της έννοιας της ασφαλούς τρίτης χώρας πρέπει να συμμορφώνεται με την ε, οδηγία για ε, τις επιστροφές και να συμμορφώνεται πλήρως με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Η Τουρκία είναι χαρακτηρισμένη ως ασφαλής χώρα για την ε, επαναπροώθηση τόσο σύρων όσο και μη σύρων των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν χαρακτηριστεί μη παραδεκτές. Και αυτό, αυτή η συμφωνία υπόκειται σε στενό έλεγχο ε, του νομοθετικού πλαισίου της Τουρκίας αλλά και έλεγχο της ε, μεταχείρισης ε, που επιφυλάσσει η Τουρκία στους πρόσφυγες, στους ετούντες άσυλο. Υπάρχει έλεγχος λοιπόν και των τουρκικών αρχών για τις περιπτώσεις αυτές επαναπρόθεσης. Όπως είπα και πριν, πάντα Εκτός από την γενική αξιολόγηση γίνεται και μια μεμονωμένη αξιολόγηση για την ασφάλεια στην Τουρκία και την ασφάλεια των ατόμων που επαναπροωθούνται. Εδώ και δύο χρόνια ισχύει αυτή η συμφωνία, εδώ και δύο χρόνια υπάρχουν αυτές οι ανταλλαγές ε, μεταξύ των ελληνικών και τουρκικών αρχών. Έχουμε δει αρκετέ περιπτώσεις ε, στις οποίες οι επιτροπές ε, ένστασης έχουν αποφανθεί ότι η Τουρκία δεν είναι ασφαλής χώρα για συγκεκριμένες περιπτώσεις ετούντων άσυλο. Και σε αρκετές περιπτώσεις οι αρχές ε, που ε, επεξεργάζονται πρώτες στην αίτηση ασύλου φτάνουν ε, στα δικαστήρια. Το Συμβούλιο της Επικρατείας στην Ελλάδα πέρυσι το Σεπτέμβριο απεφάνθη ότι η Τουρκία είναι επί της αρχής ε, μια χώρα που μπορεί να χαρακτηριστεί ως ασφαλής τρίτη χώρα. Πάντα βέβαια ε, μετά από αξιολόγηση κατά περίπτωση. Και γενικότερα σε ό,τι αφορά την Τουρκία να πω ότι είναι γνωστό πως ορισμένες πτυχές ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι πτυχές τις οποίες έχει ασκηθεί κριτική στα πλαίσια της ε, διαδικασίας προσχώρησης. Η αξιολόγηση που πρέπει να γίνει όμως ε, στην περίπτωση αυτή είναι τι συμπεριφορά θα επιφυλάσσεται στα άτομα αυτά τα οποία προσπαθούν παρά την επαναεισέλθουν στην Ελλάδα και επαναπροωθούνται στην Τουρκία. Να υπενθυμίσω επίσης ότι η Τουρκία είναι η χώρα που υποδέχεται τους περισσότερους πρόσφυγες ε, στην ε, περιοχή και το καθεστώς ε, των προσφύγων αυτών χαρακτηρίζεται από ποιοτικά πρότυπα. Η μεταχείρισή τους λοιπόν είναι καλή σε γενικέ γραμμές, έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, σε υπηρεσίες υγείας, στην αγορά εργασία και σε κοινωνικο-οικονομική στήριξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν και συνεχίζει να είναι ε, χορηγό σημαντικών ε, ποσών βοήθειας ε, στην Τουρκία μέσω της διευκόλυνσης αυτής έχουν ήδη εκταμιευθεί ποσά τα οποία μόλις λήξει το πρόγραμμα θα ανέλθουν στα περίπου 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόοδος. Ασφαλής τρίτη χώρα λοιπόν η Τουρκία ασφαλής τρίτη χώρα και ε, μάλιστα είναι αυτό περίεργο αν ε, δούμε τις αιτήσεις ασύλου που προέρχονται από την ε, Τουρκία, από Τούρκους επικούς. Τώρα όμως ο λόγος στους συναδέλφους. Κανείς δεν θέλει το λόγο. Ο κύριος Μαριάς. Κυρία Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα να επισημάνουμε ότι δεν πρόκειται για διεθνή συνθήκη Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας είναι μια δήλωση κοινή και από πλευράς νομικής βάσεως δεν έχει την έννοια της συνθήκης, της διεθνούς συνθήκης όπως την ξέρουμε. Πρόκειται για μια δήλωση. Παρά τα αυτά, να ακολουθήσουμε την ομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον παράγει ένομα αποτελέσματα, μπορεί και αυτή η δήλωση να ελεγχθεί δικαστικά και να κριθεί. Δεύτερη παρατήρηση έχουν περάσει χιλιάδες ε, πρόσφυγες και χιλιάδες παράνομοι μετανάστες στα ελληνικά νησιά από την Τουρκία. Η Τουρκία που γνωρίζουμε ότι έχει ένα ε, καθεστώς ε, αυταρχικό, αντιδημοκρατικό, δεν υπάρχουν δικαιώματα στην Τουρκία και δεν μπορεί να κυκλοφορήσει κανείς ελεύθερος αν δεν το θέλει το καθεστώς. Οπότε το ερώτημα είναι πώς περνάνε αυτές οι χιλιάδες πρόσφυγες και οι χιλιάδες παράνομοι μετανάστες στα νησιά του Αιγαίου όλους τους αντιφρονούντες ο Ερντογάν τους έχει βάλει φυλακή. Άρα λοιπόν υπάρχει ανοχή και συνενοχή και συμμετοχή του τουρκικού καθεστώτος μαζί με τους δουλέμπορους στο να γίνεται αυτή η διακίνηση, αυτή η πραγματικότητα. Και πλέον δεν έχουμε μόνο χιλιάδες πρόσφυγες και χιλιάδες παράνομους μετανάστες στα νησιά του Αιγαίου, πάνω από 20.000. Ακόμη και όταν γίνονται μετακινήσεις ε, προς την υπηρετική Ελλάδα, μόλις υπάρξει ένα κενό σε κάποιο νησί, αμέσως έρχονται με βάρκες από την άλλη πλευρά. Τώρα έχουμε και παράνομη μετακίνηση από την Τουρκία προς τη Βουλγαρία και από τη Βουλγαρία προς την Ελλάδα ή απευθείας από την Τουρκία στην Ελλάδα χερσαία. Άρα λοιπόν το πρώτο που θα πρέπει να δει και η Κομισιόν και να δούμε και εμείς είναι ότι πρέπει να υπάρξει αποφασιστικό μήνυμα στην Τουρκία διότι παίρνει και τα χρήματα δισεκατομμύρια, 6 δισεκατομμύρια θα πάρει και παίρνει για τα θέματα του προσφυγικού και παρά τα αυτά κάνει χοντρές business, αφήνει όλο τον κόσμο αυτό προφανώς πληρώνοντας λεφτά, διότι όλοι αυτοί πληρώνουν από 1.000 εως 2000 2-3.000 ευρώ ανάλογα και πάνε και περνούν στην Ελλάδα. Επομένω υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα εκμετάλλευση από τι ίδιε τι αρχέ τη Τουρκία. Διότι κανεί δεν μπορεί να κυκλοφορήσει ελεύθερο στην Τουρκία. Πώ περνάνε αυτοί απέναντι, πώ περνάνε από το Χερσαία από την Τουρκία στην Ελλάδα. Λοιπόν, Δεύτερο, υπήρχε μια απαράδεκτη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ελληνικών αρχών και της Τουρκίας όσοι πρόσφυγες είναι στα νησιά να μην μετακινούνται στην Επιρωτική Ελλάδα. Με αποτέλεσμα να μην χωράνε πλέον στα νησιά. Αυτό είναι απαράδεκτο και παράνομο και θα πρέπει να ανατραπεί. Και το πιο βασικό είναι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν θέλουν να παραμείνουν στην Ελλάδα. Ο στόχο του είναι να πάνε σε άλλε χώρε. Εδώ υπάρχει ευθύνη τη Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί σταμάτησε το πρόγραμμα μετεγκαταστάσεων. Το πρόγραμμα μετεγκαταστάσεων εκτελέστηκε και τελειώνω με αυτό. Τελειώνω. Εκτελέστηκε μόνο κατά 30% από τη Γερμανία, 25% από τη Γαλλία και υπάρχουν άλλε χώρε όπω είναι η Πολωνία, η Ουγγαρία που δεν έχουν κάνει καμία μετεγκατάσταση. Άρα λοιπόν δεν μπορεί η Ελλάδα να σηκώσει αυτό το βάρο αυτή τη κατάσταση που επικρατεί. Χρειάζονται συγκεκριμένα μέτρα. Κυρώσει κατά τη Τουρκία διότι δεν τηρεί τα συμφωνηθέντα να υπάρχει καλύτερη φύλαξη των συνόρων και να κάνει τη δουλειά της πολύ καλύτερα η Frontex και η Frontex λέει μια δικαιολογία. Ξέρετε κάτι, είναι θάλασσα, δεν μπορώ να ελέγξω. Μάλιστα. Στην ξηρά, στον Εύρο, Εκεί γιατί δεν υπάρχει σοβαρός έλεγχος. Και τρίτον, να ξαναδούμε το πρόγραμμα μετεγκαταστάσεων για να μπορούν να μετεγκατασταθούν όσοι θέλουν σε άλλες χώρες. Και τέταρτον, να πρέπει να γίνουν πιο ουσιαστικές οι διαδικασίες παροχής ασύλου και στην Ελλάδα. Δηλαδή να τηρείται το κράτος δικαίου, να τηρούνται οι προϋποθέσεις, αλλά να μην κάνουμε τρία χρόνια για να τελειώσει μια υπόθεση παροχής χορήγησης ασύλου. Νομίζω ότι εδώ πολλές φορές γίνεται κατάχρηση δικαιώματος από όσους κάνουν αίτηση. Πολλοί από αυτούς δεν δικαιούνται. Ξέρουν ότι θα περάσουν τρία χρόνια για να βγει η απόφαση, οπότε έρχονται και αν τελειώσει η υπόθεσή τους, αν κάποτε τελειώσει, αν βρεθούν, θα υποστούν, αν υποστούν συνέπειες που δεν υφίστανται καμία συνέπεια. Άρα λοιπόν είναι πολλά τα θέματα που πρέπει να δούμε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Thank you very much. Well, interesting discussion, but this is ενδιαφέρουσα η συζήτηση αυτή, αλλά δεν αφορά αυτήν ακριβώ την αναφορά. Θα ήθελα να συγκεντρώσουμε τα σχόλιά μα σε αυτή την αναφορά, αν είναι δυνατόν. Να συνοψίσω. Α, ο κύριος Ζαριανόπουλο. Παρακαλώ πολύ σύντομα να είστε κύριε Ζαριανόπουλε. Γιατί είμαστε πίσω, σε μισή ώρα πίσω. Η, ε, πρόκειται περί δήλωση μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Τουρκία. Ανεξάρτητα από τη νομική τη μορφή, λειτουργεί σαν συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση και Τουρκία και με τη συμφωνία της ελληνικής κυβέρνησης και μάλιστα μια συμφωνία σκληρότατης και απαράδεκτης. Είναι αυτή η οποία είναι υπεύθυνη για τον εγκλωβισμό χιλιάδων στα ελληνικά νησιά δίπλα από την Τουρκία σε απαράδεκτες συνθήκες, όλοι το ξέρετε. Που βεβαίως δεν μπορούν να μετακινηθούν ούτε καν προς την υπηρετική Ελλάδα. Είναι παραβίαση της συνθήκης της Γενέβης, σαφέστατη, για τους πρόσφυγες και βεβαίω εδώ επάνω δημιουργούνται και διάφορα ζητήματα. Παράδειγμα το ερώτημα αν η Τουρκία είναι ασφαλή χώρα. Αποδεικνύεται κατά την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η Τουρκία είναι ασφαλή χώρα à la carte. Άλλε φορέ είναι και άλλε φορέ δεν είναι. Είναι αποτέλεσμα παζαριών πολιτικών αυτό που γίνεται. Προωθείται και μέσω τη οδηγία του Δουβλίνου η παραμονή στην πρώτη χώρα, στην πρώτη χώρα εισόδου. Εδώ έχουμε μιλάμε για το πρώτο νησί εισόδου στην Ελλάδα, σε απαράδεκτε συνθήκε. Και βεβαίω, για να τελειώσω με αυτό, υπάρχει και ένας διαχωρισμός που γίνεται που μπορεί στην νομική επιστήμη να έχει κάποια ουσία αλλά στην πραγματικότητα πολλές φορές είναι επικίνδυνος. Δηλαδή πρόσφυγα στον πόλεμο στις συνθήκες που, που λέμε. Αυτό το παράνομος μετανάστης τι ακριβώς είναι που πρέπει να ξαναγυρίσει πίσω. Στην πραγματικότητα είναι αυτός ο οποίος μετά από τον πόλεμο δεν έχει πηγές να ζήσει στη χώρα του την κατεστραμμένη και γίνεται παράνομος μετανάστης. Έρχεται από την Αφρική όπου δεν μπορεί να ζήσει. Αυτού του είδου οι διαχωρισμοί στην πραγματικότητα ενισχύουν ακροδεξιέ απόψει. Και στην Ελλάδα και στην Ιταλία και σε, και σε όλο το τέτοιο. Αυτά λοιπόν πρέπει να σταματήσουν και να πάμε στην ουσία. Πρώτον, ποια είναι η αιτία, η παραγωγός αιτία των προσφύγων ο πόλεμο που συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση πρώτον. Και δεύτερον, ποια είναι η στάση τη απέναντι στου πρόσφυγε. Απαράδεκτη. Αυτή η συμφωνία με την Τουρκία πρέπει να σταματήσει και να ισχύσει η συνθήκη τη Γενέβη. Thank Όπως είπα, θέλω να εστιάσουμε σε αυτή την αναφορά και κανείς δεν μου έκανε μια πρόταση. Όλοι γνωρίζουμε περί τίνος πρόκειται. Νομίζω ότι εξαντλήσαμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Ακούσαμε την Άντζελα, και από άλλους ερωτήσεις προς την Κομισιόν. Έχουμε κάνει ό,τι μπορούσαμε. Νομίζω ότι είναι ώρα να κλείσουμε αυτήν την αναφορά. Δεν έχουμε να εξετάσουμε τίποτα άλλο. Έχουμε την οδηγία υποβοήθησης που πρέπει πραγματικά να προσπαθήσουμε να βγάλουμε κάποιο αποτέλεσμα, αλλά δεν νομίζω ότι αυτή την αναφορά χρειάζεται να την κρατήσουμε ανοιχτή. Εντάξει, ωραία υπόθεση. και επειδή είναι μεγάλο πολιτικό ζήτημα, εγώ από την πλευρά μου δεν θα συμφωνήσω να κλείσει. Είναι μεγάλο πολιτικό ζήτημα, θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτό. Yeah. Yeah. But listen, we have done what we... Ωραία. Όμω κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Υπάρχουν και άλλε αναφορέ για το ίδιο θέμα. Και η οδηγία είναι πολύ πιο σημαντική. Εδώ θα πρέπει να πούμε στον αναφέροντα ότι εξαντλήσαμε τι δυνατότητέ μα. Και νομίζω ότι οι συνάδελφοι συμφωνούν μπορούμε να κλείσουμε αυτή την αναφορά. Κύριε Μαριά. Θα να ακούσω την πρότασή σας. Η δικιά μας πρόταση ως CCR είναι η εξή. Πρώτον, θα πρέπει να αποσταλεί η αναφορά αυτή στην Επιτροπή Εξωτερικών, διότι αυτό το θέμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό. Δεύτερον, να ζητήσουμε από την Κομισιόν να εξετάσει αρμοδίως ε, πώς μπορεί να προετοιμάσει η Κομισιόν πρόταση για επιβολή κυρώσεων κατά της Τουρκίας. Και τρίτον, αυτή η αναφορά πρέπει να μείνει ανοιχτή για τον εξή λόγο. Γιατί αυτή είναι η αιτία όλων των άλλων αναφορών για τις οποίες συζητούμε γύρω από το προσφυγικό μεταναστευτικό στην Ελλάδα. Αυτή είναι η βάση. Αν αλλάξει η βάση, προφανώς θα έχουμε άλλες συνθήκες. Αν παραμείνει αυτή η βάση, θα έχουμε όλες αυτές τις αναφορές και άλλες που θα έρθουν. Επομένως, δεν μπορεί να κλείσει αυτή η αναφορά, γιατί είναι the basis όλου του θέματος το οποίο συζητούμε. Okay. I just need... Ωραία. Να σας πω ότι η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων δεν έχει να κάνει τίποτα με αυτή τη δήλωση. Η δήλωση είναι μεταξύ αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. στο Συμβούλιο αρχή, Αρχηγοί Κρατών Κυβερνήσεων έκλεισαν αυτό που ήταν στην αρχή μια συμφωνία. Συμφωνία το είπα στην αρχή, μετά η νομική υπηρεσία που δεν είναι συμφωνία, γιατί μετά κάποιο ε, μπορεί να προσφύγει στο κοινοβούλιο, ε, στο δικαστήριο, επειδή παρακάμφθηκε το κοινοβούλιο. Οπότε το ονόμασαν διαφορετικά. Πρόκειται λοιπόν για δήλωση. Ωραία. Για αυτή τη δήλωση το κοινοβούλιο δεν έχει καμία αρμοδιότητα. Ευκαιρία να πάρουμε την μπάλα στο γήπεδό μας. Όχι, μην είμαστε αφελείς, μην είμαστε αφελείς. Ξέρουμε περί τίνο πρόκειται. Και το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να κλείσουμε αυτήν την αναφορά. Νομίζω ότι έχω τη στήριξη των συνάδελφων, έτσι. να διευκονίσω ότι η θέση μας ήταν η πρόταση συγκεκριμένη που σας ανέφερα, εντάξει. Ωραία. ECR διαφέρει ακόμα και σήμερα πολύ συχνά. Ωραία, περνάμε στην επόμενη αναφορά. Η 75 εκ μέρου τη Οργάνωση Παγκόσμια Ομοσπονδία Συνδικάτων σχετικά με τη δύσκολη κατάσταση που βρίσκονται οι διακινούμενοι εργαζόμενοι στη Φότζια τη Ιταλία και την 374 του συναδέλφου κυρίου Ζαριανόπουλου. Μέτρα, λήψη άμεσων μέτρων για την προστασία Α, όχι, μπερδεύτηκα, πέρασα μία. Σο, βέβαια, συγγνώμη. Συγγνώμη, είμαστε στο 20 της ημερήσιας διάταξης. Έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ πραγματικά. Αναφορά υπαρθμών 620 και αναφορά υπαρθμών 225. Ο κ. Φαρμάκης είναι ο αναφέρον. Σας δίνω το λόγο για 5 λεπτά. Ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε, και τα υπόλοιπα μέλη που δεχτήκατε να συζητήσουμε την αναφορά μας. Η Όλαφ αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή τη στιγμή ερευνά στην Ελλάδα με βάση τα πορίσματα που έχει αναφέρει η αναφορά μας. Εδώ και 21 χρόνια δραστηριοποιούμε στην ελληνική κοινωνία των πολιτών και πιστεύουμε ότι αυτά τα έγγραφα, όπως και άλλα έγγραφα που υποβάλαμε πρόσφατα, έχουν αποδείξει την αποτυχία του ελληνικού κράτους να τηρήσει τις διεθνείς της και τις εθνικές και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της να εξασφαλίσει αξιοπρεπείς συνθήκες υποδοχής των ετούντων. Βλέπετε μία φωτογραφία, δεν σας δείξω καμία άλλη. Νομίζω ότι είναι πολύ γλαφυρή ε, έχουμε ρεπορτάζ στις εφημερίδες καθημερινά πριν από δύο εβδομάδες ε, ο Επίτροπος Συμβουλίου της Ευρώπης έκανε πολύ σκληρά σχόλια για τις συνθήκες που επικρατούν στη Λέσβο και τη Σάμο κυρίως αλλά και στα υπόλοιπα ελληνικά νησιά. Το ελληνικό κράτος λοιπόν απέτυχε να εξασφαλίσει αξιοπρεπείς συνθήκες υποδοχής ε, στους ετούντες διεθνή προστασία και επίσης απέτυχε να εφαρμόσει να χρησιμοποιήσει σωστά τα 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ που χορηγήθηκαν στην Ελλάδα. Το έχουμε αναφέρει στην αναφορά μας. Τα, το, μεγαλύτερο από αυτά, το μεγαλύτερο τμήμα αυτού του ποσού απορροφήθηκε, αλλά ε, είδαμε πολλές καταχρήσεις ε, στις ε, πολιτικές ε, συμβάσεων. Μια πρόσφατη έρευνα για θέματα catering, για παράδειγμα, έδωσε αυτά τα αποτελέσματα. Έχουμε στοιχεία ε, τουλάχιστον αδιαφάνειας, αλλά, σίγου, αλλά και κατάχρησης. Μιλάμε για τις δραστηριότητες catering και κατασκευής προκατασκευασμένων, εγκατάστασης προκατασκευασμένων οικειών. Επίσης, το ελληνικό κράτος απέτυχε να διασφαλίσει την εφαρμογή των κανόνων δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως αυτές έχουν μεταγραφεί στο ελληνικό δίκαιο. Προτείνουμε να μείνει ανοιχτή η αναφορά προκειμένου να διερευνηθεί περαιτέρω. Προτείνουμε επίσης η Επιτροπή σα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γέννη να δημιουργήσουν, να, να, μια επίσκεψη στην Ελλάδα Έρευνα, διερευνητική επισκέψη, αναμένοντας ε, βέβαια πρώτα την επιτυχή ολοκλήρωση των ασιών της Όλαφ που ελπίζουμε ότι θα τελειώσουν γρήγορα και θα δημοσιευθούν τα αποτελέσματα σύντομα. Όπως ε, γνωρίζετε ο συνολικός αριθμός ε, των ετούντων άσυλων στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν 65.000 άτομα, σημαντικό νούμερο αλλά δεν έχει προφανώς καμία αναλογικότητα με τα 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία έχουν χορηγηθεί στην Ελλάδα συνολικά. Επίσης, ε, η, ε, να αναγνωρίσω το έργο της κυρίας Ελένης Τάκου, της Μαρίας Παρασκευά, της Ελένης Παπαδοπούλου που δεν είναι μαζί μας σήμερα. Καθώς επίσης και θα δώσω το λόγο και στην συνάδελφό μου την Ατάσα για να ολοκληρώσουμε μερικές φράσεις. Οι αιτούντε άσυλο όταν φτάνουν στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν μια κατάσταση που έλλειψη χώρου, ε, πολύ κακές και ανασφαλείς συνθήκες ε, στην υποδοχή. Αυτό οδήγησε συχνά στην Ελλάδα σε παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε απώλεια ζωής. Ε, η αρμοστία για τους πρόσφυγες έχει καταγγείλει αυτές τις συνθήκες. Ε, το ίδιο το ελληνικό κράτος έχει δεχτεί ε, τις αδυναμίες. Υπάρχει ανυπαρξία κυβέρνησης επιτόπου. Πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ έχουν, έχει δοθεί για να βοηθηθεί η ελληνική κυβέρνηση να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το Κοινοβούλιο πάντοτε λέει ότι η χρηματοδότηση τη Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να παρακολουθείτε προκειμένου να χρησιμοποιείται με τρόπο που θα κάνει σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τι διεθνεί προδιαγραφέ. Ε, πολύ μεγάλη κακοδιαχείριση στην Ελλάδα. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα ληφθούν μέτρα διότι απειλούνται ζωέ. Το Κοινοβούλιο γνωρίζει πολύ καλά ότι οι συνθήκε υποδοχή στην Ελλάδα ε, είναι πολύ προβληματικές. Η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες το αναφέρει επίσης. Θα πρέπει η απουσία δράσης να μην γίνει συνενοχή. Όλοι γνωρίζουμε πως ε, είμαστε όλοι ίσοι και έχουμε δικαίωμα στην αξιοπρέπειά μας. Ζητάμε τη συνεργασία σας. Σα ευχαριστώ. Θα δώσουμε τώρα το λόγο απευθείας στην ε, εκπρόσωπο της Κομισιόν, την κυρία Τουρλουμούση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις που υποβάλαμε προς την Επιτροπή σας και σύμφωνα και με τα στοιχεία που υπέβαλαν οι αναφέροντες και τους οποίους ευχαριστώ για τη συνεισφορά, θα ήθελα να πω ότι η Κομισιόν εξακολουθεί να παρακολουθεί στενά την κατάσταση στην Ελλάδα. Είναι γνωστό ότι από το 2015 όπου η μεταναστευτική κρίση ξεκίνησε η Κομισιόν υποστηρίζει την Ελλάδα επιχειρησιακά και χρηματοδοτικά. Όπως λέγεται εδώ κατά τις πληροφορίες της αρχής μας υποβολής προς την Επιτροπή σας η ΓΔ Home, ΕΚΟ, η SRSS και άλλοι ευρωπαϊκοί οργανισμοί και γραφεία υποστήριξης, η Frontex, η Europol συνεχώς υποστήριξαν την Ελλάδα σε επιχειρησιακό επίπεδο προκειμένου να βοηθήσουν τις ελληνικές αρχές να ανταπεξέλθουν προς την κρίση. Πέρασε χρόνος η μεταναστευτική εισρωή δεν είναι τόσο έντονη όσο ήταν στο παρελθόν. Ωστόσο, την κατάσταση θα πρέπει να παρακολουθούμε στενά και η υποστήριξη από πλευράς κομισιών και λοιπόν φορέων θα πρέπει να συνεχιστεί. Εξού και έχουν αναπτυχθεί ομάδες από την ΓΔ Home και ΕΚΟ στο έδαφος, εμπειρογνώμονες, προσωρινό προσωπικό και από άλλους οργανισμούς για να βοηθηθούν οι ελληνικές αρχές να συμπληρώσουν τις επιχειρησιακές τους δυνατότητες αλλά και να τους βοηθήσουμε να εγκαταστήσουν βιώσιμες και επαρκείς πολιτικές ασύλου και ιδιαίτερα υποδοχής γιατί αυτή είναι και η ουσία της αναφοράς. Έγιναν κάποια πράγματα, έχει αυξηθεί το δυναμικό υποδοχής, ιδιαίτερα στην εδωχώρα. Έχει γίνει μια χρηματοδότηση προγράμματος οικιστικού και με την συνεπικουρία και άλλων οργανώσεων με 25 συνολικά 27 συνολικά χιλιάδες ε, θέσεις. Και δόθη και η νομικά απαραίτητη ενίσχυση για τους ετούντες άσυλο. Υπάρχει μια συνεχιζόμενη προσπάθεια βελτίωση των προτύπων, ιδιαίτερα για μέλη ευάλωτων ομάδων και ασυνόδευτους ανηλίκους. Εδώ πρέπει να πούμε ότι η Κομισιόν διαρκώς και σε όλα τα επίπεδα ενημέρωνε και ειδοποιούσε τις ελληνικές αρχές μέσω τεχνικών επισκέψεων και άλλων επισκέψεων και όχι μόνο μέσω της βοήθειας επιτόπου για τα προβλήματα που ακόμα παραμένουν και τα οποία πρέπει άμεσα να, να επιληθούν. Και ως πρόσθετο σημείο της δικής μας υποβολής καθότι αναφερόμαστε στην, στις χρηματοδοτικές προβλέψεις για 17 θα συνεχιστούν 18 και 19 προκειμένου να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τις ελληνικές αρχές για να επικαιροποιήσουν και να βελτιώσουν την πολιτική τους υποδοχής επί τη βάση πλήρων και υγιών στατιστικών δεδομένων και επί τη βάση των απαραίτητων υπηρεσιών που θα πρέπει να παρέχονται. Όπως έλεγα, εξακολουθούμε να παρακολουθούμε στενά την κατάσταση, διότι ο ρόλος της Κομισιόν είναι να διασφαλίζει ότι θα υπάρχουν επαρκείς συνθήκες υποδοχής στους ανθρώπους που έχουν δικαίωμα πρόσβαση σε αυτές. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Τώρα το λόγο έχουν τα μέλη. Η κυρία Σακοράφα πρώτα απ' όλα. Ε, να είμαι σαφή, λέει η πρόεδρο. ένα λεπτό σας παρακαλώ, όχι παραπάνω, θα το μετρήσω γιατί έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη έτσι και αλλιώ, γιατί πρέπει να φύγω και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Θα πρέπει να πάω στην ΑΦΕΤ. Εδώ βλέπουμε σήμερα ότι έχουμε σοβαρέ καταγγελίε από του αναφέροντε, καταγγελίε οι οποίε επιβεβαιώνονται και από δημοσιεύματα του τύπου στην, ε, στη χώρα μα. Ε, ε, δημοσιεύματα όσον αφορά την κακοδιαχείριση των κοινωτικών πόρων, κυρίω του Ταμείου Ασύλου, τη μετανάστευση και τη ένταξη και του Ταμείου Εσωτερική Ασφάλειας και Μηχανισμού έκτακτη υποστηρίξη, πράγμα το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα την αποτυχία τη χώρα να εκπληρώσει τις διεθνείς ευρωπαϊκές ε, και εθνικέ υποχρεώσει σχετικά με την καθιέρωση των ανθρωπίνων αξιοπρεπών και ανθρώπινων συνθήκων διαβίωση των ετούντων άσυλο στην χώρα. Κυρία Πρόεδρε, είναι γεγονό ότι κλήθηκε η Ελλάδα να σηκώσει ένα βάρο δυσανάλογο σε σχέση και με το μέγεθό τη, αλλά και με το μέγεθο τη κρίση που περνάει αυτή τη στιγμή. Όμω αυτό δεν έχει καμιά δικαιολογία, διότι εδώ μιλάμε για ανθρώπινε ζωέ. Μιλάμε για ανθρώπινε ζωέ, οι οποίε κατέληξαν, θα έλεγα, μετά από τραγικέ διαδικασίε σε αυτή τη χώρα, που, κλήθηκαν, που κλήθηκε η Ελλάδα μέσα από συμφωνίες να διεκπαιρεώσει ε, την, την υποστήριξή τους και αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο έλεος του Θεού. Θεωρώ ότι έχουμε υποχρέωση να κρατήσουμε ανοιχτή τη συγκεκριμένη ε, αναφορά. Ε, ε, πρέπει να σταλεί στην Ελλάδα μήνυμα ότι θα πρέπει να δώσει οποιαδήποτε στοιχεία που να αφορούν στην διαχείριση αυτών των κονδυλίων, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ακριβώ επειδή τα δημοσιεύματα δεν αφορούν μόνο την κακοδιαχείριση από την πλευρά τη χώρα, από την πλευρά τη κυβέρνηση και αφορούν και στις, σε κάποιε, όχι όλε για να είμαστε ε, ε, καθαρή ε, ΜΚΟ οι οποίες δραστηριοποιούνται στην περιοχή θα πρέπει ο έλεγχος να είναι πλήρης και ενδελεχής προς κάθε κατεύθυνση. Αυτά και ευχαριστώ πολύ. Thank Σας ευχαριστώ κύριε Μαριάς. Κυρία Πρόεδρε, να ευχαριστήσω τους αναφέροντες. Με αυτά που λένε επιβεβαιώνουν αυτά τα οποία καταγγέλω στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το Σεπτέμβριο του 2015 είχα πει ότι γίνεται ένα μεγάλο πάρτι και το πάρτι αυτό το κάνουν πάρα πολλέ ΜΚΟ, οι οποίε είναι ανεξέλεγκτε. Διότι τα κονδύλια τη Ευρωπαϊκή Ένωση, το 1,6 δι που ακούσαμε, από αυτά 460 εκατομμύρια ευρώ πηγαίνουν απευθεία από την Κομισιόν σε μη κυβερνητικέ οργανώσει, εκ των οποίων με βάση αυτά που μα είπε ο κ. Τηλιανίδης πρόσφατα, 410 εκατομμύρια ευρώ έχουν συμβολεοποιηθεί, δηλαδή έχουν ξεκινήσει διαδικασίε. Επ' αυτών λοιπόν έχουν γίνει καταγγελίες και θα πρέπει η Όλαφ να επεκτείνει τον έλεγχό τη και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Ορισμένε από αυτές είναι πλέον κράτος εν κράτη. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δει η Κομισιόν γιατί έχει ευθύνη. Δεύτερον, είχαμε πει ότι τα κονδύλια πρέπει να μην πηγαίνουν στι μη κυβερνητικέ οργανώσει, να πάνε στην τοπική αυτοδιοίκηση και στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση που υφίσταται το τεράστιο βάρο και η οποία πρέπει να πάρει μέτρα και η οποία πληρώνει αυτή τη στιγμή δικά τη κονδύλια και όπου υπάρχουν καλύτερε διαδικασίε. Επιπλέον, υπάρχει και πρέπει να γίνει έλεγχο από πλευρά τη Όλαφ και στις κρατικές υπηρεσίες της Ελλάδος. Αυτό που αναφέρθηκε για τα γεύματα είναι σκανδαλώδες. Το έχω καταγγείλει δέκα φορές στην Ολομέλεια. Δηλαδή, παρασκευάζονται τα γεύματα στην Κόρινθο. Από την Κόρινθο πηγαίνουν στον Πειραιά. Από τον Πειραιά με καράβι στη Σάμο και στη Σάμο θερμαίνονται για να τα φάνε οι πρόσφυγες. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που ευθύνεται η Κομισιόν γιατί το έχω πει πριν τρία χρόνια και έκλεινε τα μάτια. Και τώρα που έσκασε όλη αυτή η ιστορία έρχεται η Κομισιόν να πει τι θα κάνει. Να μπει η Όλαφ να ελέγξει όλα αυτά τα πράγματα. Του Τους τα έχουμε πει εδώ και χρόνια. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Μπορώ αυτό να σας πω ότι η Όλαφ αυτή τη στιγμή ερευνά τις καταγγελίες σχετικά με την παροχή ε, διατροφής, τροφίμων, εν στους ε, πρόσφυγες. Πρέπει να το λάβουμε πόσο πολύ σοβαρά. Η κυρία Κούνεβα. Η Ελλάδα, ενώ δεν υπήρξε ποτέ χώρα υποδοχή προσφύγων, κατάφερε σε πάρα πολύ σύντομο ιστορικά διάστημα να φτιάξει δομέ για πάνω από 60.000 ανθρώπου, του οποίου έπρεπε να στεγάσει, να τρέψει και να περιθάψει. Ήταν άθλος αυτό που καταφέραμε. Η ευρωπαϊκή οικονομική βοήθεια πηγαίνει τόσο στο κρατικό προπολογισμό όσο και στι μη κυβερνητικέ οργανώσει. Και οποιαδήποτε ανταπάνη κάνει η κυβέρνηση δημοσιεύεται υποχρεωτικά. Υπάρχει διάβγεια σε αυτό. Αντιθέτω, και ενώ οι αρμόδιοι υπουργοί έχουν ζητήσει τουλάχιστον τέσσερι φορέ στη Βουλή να παρουσιάζουν και οι μη κυβερνητικέ οργανώσει μηνιαίω τι δαπάνε του, αρνιούνται συστηματικά να το κάνουν. Είναι οι συνθήκε. Όχι. Προσπαθούμε όμω συνεχώ να βελτιώνουμε απέναντι σε αριθμού που κάνουν τι υπηρεσίε να λυγίζουν. Έχουμε, έχουν έρθει Ωραία. Αυτή τη στιγμή γίνεται έρευνα από το Όλαφ στην Ελλάδα και δεν έχει βρεθεί κάτι σχετικά με τα κοντήλια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ζαριανόπουλος. Ένα λεπτό παρακαλώ. Τυχαία σημαίνει λάθος και εδώ δεν πρόκειται για λάθος, είναι για συνειδητή πολιτική. Δεν θέλω να μπω στα ζητήματα των ερευνών που γίνονται και πρέπει να γίνονται για να διαπιστωθούν οι όποιες παραβιάσεις έχουν γίνει και στο κράτος και στις ΜΚΟ κτλ. Βεβαίω η κατάσταση είναι απαράδεκτη. Και γιατί είναι απαράδεκτη, διότι μέσα στο ζήτημα διαχείρισης του προσφυγικού ζητήματος μπαίνουν ιδιωτικά επιχειρηματικά συμφέροντα και το εκμεταλλεύονται για κέρδη και βεβαίως τα με περισσότερα κονδύλια, συντριπτικά περισσότερα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείριση του προσφυγικού τα παίρνουν οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις, οι ΜΚΟ, άλλο πάρτι, πάρτι κυριολεκτικά, που δεν δίνουν και στοιχεία. Με αυτή την άποψη το ζήτημα δεν είναι ο έλεγχος. Το ζήτημα είναι ο αποκλεισμό των μη κυβερνητικών οργανώσεων από τη διαχείριση του προσφυγικού. Δεν έχουν καμία δουλειά. Η αποκλειστική ευθύνη του κράτους και όλων των κρατών για το προσφυγικό ζήτημα και βεβαίω η συνέχιση του ελέγχου από τις δικαστικές αρχές της χώρα για όλα αυτά τα ζητήματα. Με αυτή την έννοια να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά. Σα ευχαριστώ πολύ. Έχουμε ζητήσει γνωμοδότηση από την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ Πολιτικών Ελευθερινιών. και η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ λοιπόν είναι της άποψης ότι η, η χρήση των κονδυλίων είναι μια περιοχή για την οποία υπάρχουν ελάχιστες πληροφορίες και μάλιστα τα ποσοστά απορρόφησης του MMISF από τις ελληνικές αρχές παραμένουν πάρα πολύ χαμηλά. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε για να ολοκληρώσουμε με το θέμα, να κρατήσουμε ανοιχτή την αναφορά και να περιμένουμε το πόρισμα της έρευνας της Όλαφ, να γράψουμε στις ελληνικές αρχές και να εκφράσουμε την ε, έντονη ανησυχία μας για τις συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων, όχι μόνο στα νησιά αλλά και στην ενδοχώρα και να ζητήσουμε λεπτομέρειες για την ε, χρήση των ε, κονδυλίων που έχουν εκταμιευθεί. Προβλέπουμε λοιπόν ε, εξελίξεις γρήγορα. Ωραία. Τώρα, ο κύριος Αργιανόπουλος ήρθε η σειρά σας μία ώρα αργότερα από την προγραμματισμένη. Δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε. Έχουμε την αναφορά 75 του 2018 και 374 του 2018. Έχετε 2,5 λεπτά έκαστος. Νομίζω φτάνει ο χρόνος διότι γνωρίζουμε το θέμα. Σας παρακαλώ να είστε περιεκτικοί ε, και να συνεργαστείτε. Και οι δύο αναφέροντες. Θα μιλήσει, ε, να το ξεκαθαρίσω, θα μιλήσει και ο εκπρόσωπος των εργατών γης, έτσι. Λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, ε, στις 9 Φεβρουαρίου αυτού του χρόνου ε, σε συνεργασία με την Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία επισκέφθηκα το γκέτο των εργατών γη στη Φότζια της Ιταλίας μία από τις μεγαλύτερες γεωγραφικές περιοχές της Ευρώπης. Δεν πρόκειται για ένα νέο πρόβλημα ούτε προσωρινό. Είναι ένα πρόβλημα πάνω από 20 χρόνια. Υπάρχουν άνθρωποι, εργάτες γης, άνδρες και γυναίκες και παιδιά, που ζουν στις συνθήκε που βλέπετε στις φωτογραφίες. Η απόλυτη βαρβαρότητα στο κέντρο της Ευρώπης, σε μια από τις πιο πλούσιες περιοχές. Δεν έχουν σπίτι, δεν έχουν ηλεκτρικό, δεν έχουν θέρμαση, δεν έχουν τις περισσότερες φορές νερό που οι θελημένα τους το κόβουν για να τους εκβιάσουν με απέλαση οι μεγάλοι κτηματίες στους οποίους δουλεύουν οι εργάτες γης. Η κατάσταση είναι απαράδεκτη και μιλάμε για πολλές γυναίκες και για παιδιά επίσης. Δεύτερον, δεν έχουν συμβόλαια. Δουλεύουν για ψίχουλα όποτε τους χρειάζονται. Τον υπόλοιπο καιρό εκβιάζονται με κάθε τρόπο από τους κτηματίες και το Ιταλικό κράτος με απέλαση για να μην ξεσηκωθούν. Μετά από λίγους μήνες τους ξαναπήρνουν στη δουλειά, χωρίς κανένα απολύτως δικαίωμα. Και για ποια περιοχή μιλάμε, για την περιοχή αγροτικής παραγωγής, μια από τις περιοχές στην Ιταλία, που το, στο πρόγραμμα του 2014-2020 η αγροτική της παραγωγή επιδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση με 1,6 δισεκατομμύρια. Πού πήγαν αυτά, σε αυτές τις συνθήκες που βλέπετε, σε αυτούς τους μισθούς που σας λέμε. Πρόκειται για βαρβαρότητα. Ανάλογες περιπτώσεις υπάρχουν και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Και έχει ξανασχοληθεί η Επιτροπή όπως για παράδειγμα με τους εργάτες γης στη Μανολάδα της Πελοποννήσου, στην παραγωγή φράολας, που έχουν χτυπηθεί ακόμα και με όπλα από τους εργοδότες. Όπως και στην Ιταλία, στα γκέτο που βλέπετε. Λίγο μετά την επίσκεψή μου δολοφονήθηκε εργάτης γης από ανθρώπους που ακόμη μένουν άγνωστοι για την Ιταλική αστυνομία. Και άλλοι 20 αυτή τη χρονιά δολοφονήθηκαν. Κλείνω με την πρόταση. Αφενός μεν βεβαίως να παραμείνει ανοιχτή Δεύτερον, να συνεχιστεί η έρευνα για όλη αυτή την κατάσταση, να σταλεί επιστολή στην Ιταλική κυβέρνηση, η οποία θα αναζητά εξηγήσει, θα αναζητά ευθύνε και να παρθούν άμεσα μέτρα για τον οικισμό, για τα ζητήματα υγείας, για τα ζητήματα περίθαλψης, για τα ζητήματα των συμβολέων εργασίας και της παραμονής τους της νόμιμης των εργατών γης στην Ιταλία ή όπου ζούνε. Άλλωστε, αγαπητές ε, κυρίες και κύριοι, από τα χέρια του τρώμε και βρισκόμαστε εδώ. Νομίζω ότι περισσότερα θα μπορέσει να σας δώσει ο εκπρόσωπος των εργατών γης δίπλα μου. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ που τηρήσατε το χρόνο ομιλίας. Κύριε Κόντε, έχετε το λόγο και θα σας ακούσουμε για τρία λεπτά. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Για μένα η παρουσία μου εδώ είναι μια ευκαιρία να δώσουμε φωνή σε αφανείς ανθρώπους, άνθρωποι που υπάρχουν, που όμως ε, είναι αφωνοί. Εδώ και πολλά χρόνια ε, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Συνδικάτων είναι δίπλα στους εργάτες γης και προσπαθεί να προασπιστεί τα δικαιώματά μας. Η γεωργία, ακόμα και στην Ιταλία, είναι ένας ε, κλάδος πολύ ανεπτυγμένος. Είναι δεύτερος παραγωγός του ελαιολάδου, στο κρασί, στα μήλα, ε, έβδομη στο καλαμπόκι, δέκατη τέταρτη παραγωγός χώρα στον κόσμο στο σιτάρι, με κύκλο ρασιών 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Ε, το, οι εξαγωγές είναι 525 εκατομμύρια ευρώ. 8% των συνολικών εξαγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή. Επίσης υπάρχει και η αγροτροφημική βιομηχανία με κέρδη πάνω από 27 δισεκατομμύρια το χρόνο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ενεκτικού Συνεδρίου της Ιταλίας, κατά τη διάρκεια της περίοδου 2014-2020, τα ε, 41,5 δισεκατομμύρια δολάρια ήταν οι επιδοτήσεις. Συν 10,5 δισεκατομμύρια από εθνικά κονδύλια. Όλα αυτά πηγαίνουν σε γεωργικές περιοχές. Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι τα άτομα που εργάζονται δεν λαμβάνουν αυτά τα ποσά. Σήμερα στην Ιταλία η εκμετάλλευση εκτείνεται σε όλη την επικράτεια. Από τον νότο μέχρι τον βορρά. Στην Ιταλία οι σχέσεις, οι σχέσεις διέπονται από ε, συμβάσεις εργασίας εθνικές, σε εθνικό επίπεδο. Στον τομέα της γεωργίας προβλέπονται ε, μισθή, ε, μεταφορά, αναγνώριση κινδύνου δικαιώματα μητρότητας, πατρότητας, ε, αναγνώριση της ανεργίας, δηλαδή επιδόματα ανεργίας κλπ. Στην πράξη όμως τι συμβαίνει. Έχουμε 400-430.000 εργάτες γης οι οποίοι ε, βρίσκονται σε κατάσταση κινδύνου. 132.000 ε, ζουν σε άθλιες συνθήκες, πάνω από 100.000 το 30% περίπου δηλαδή του συνόλου ε, εργάζονται για λιγότερο 50 μέρες το χρόνο. Αντιλαμβάνεστε γιατί μιλάμε. Μεταξύ αυτών, πολλοί είναι αλλοδαποί, μετανάστες, οι οποίοι θεωρούνται βασικό ατού της Ιταλίας λόγω του χαμηλού κόστους τους ζουν στους αγρούς, μακριά από τις πόλεις, χωρίς νερό, χωρίς ηλεκτρισμό. Βλέπετε τις φωτογραφίες, καλύβε. Εμείς εδώ όλοι φάγαμε, έχουμε σπίτια, είμαστε εδώ, αλλά μέσα στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια έχουμε ανθρώπου που ζουν σε τέτοιε συνθήκες. Αν δείτε τις φωτογραφίες, καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση βρίσκονται άνθρωποι. Δεν, είναι, δεν μπορεί καν να του θεωρήσει ανθρώπους σε, σε αυτές τις συνθήκες. Τι θέλουμε. Θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση με κάποιο τρόπο να αντιδράσει. Στην ουσία που έχει σχέση με την κοινή αγροτική πολιτική είναι ένα θέμα που έχει σχέση με την κοινή αγροτική πολιτική. Οι επιχειρήσει αυτέ χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ίδιες αυτέ οι επιχειρήσει που χρηματοδοτούνται δεν δίνουν δικαιώματα στου εργαζόμενου του. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η τροφή, το φαΐ, αποτελεί τμήμα της ταυτότητάς μας. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να απαρνηθούμε μας, δω, μας δίνει ζωή. Αλλά δεν είναι δυνατόν η ίδια η γεωργία που παράγει την τροφή να μας καταντά σκλάβους. Εμείς οι καταναλωτές θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη το πώς παράγει την τροφή την οποία καταναλώνουμε. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τις ανισότητες. Η τροφή δεν θα πρέπει να σκοτώνει, δεν είναι δυνατόν να κάνει διακρίσεις θα πρέπει να φέρνει χαρά και απόλαυση στους ανθρώπους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήσασταν σαφείς και οι δύο και βλέπω πως έχετε μεγάλη στήριξη στην αίθουσα. Να μην έχετε καμία αμφιβολία για τη στήριξη αυτή. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Εμμανουέλ Καμπό, εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επίγνωση της ε, δραματικής κατάστασης στο Ρινιάνο και στην περιοχή της Πούλια στην Ιταλία ε, και την κατάσταση των αλλοδαπών εργατών ε, γης και των συστημάτων που χρησιμοποιούνται εκεί, καθώς και έχει επίγνωση της εκμετάλλευσης χιλιάδων αλλοδαπών εργατών. Η καταπολέμηση της ε, παράνομης εργασίας και της εκμετάλλευσης ε, συμπεριλαμβανομένης αυτής των αλλοδαπών εργατών είναι μία από τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, σύμφωνα με τις ε, πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, υπόθεση αφορά και τους αλλοδαπούς εργάτες που είναι νόμιμα στην ε, επικράτεια της Ένωσης αλλά και εκείνους που δεν βρίσκονται νόμιμα σε έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η οδηγία για την νόμιμη μεταμνάστευση είναι ε, μια οδηγία που εφαρμόζεται στην περίπτωση αυτή. Όλοι οι εργάτες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ίσα και να έχουν στέγαση η οποία θα πληρεί ε, όλες τις προϋποθέσεις και θα είναι αξιοπρεπής. Θα πρέπει επίσης να υπάρχουν οι κατάλληλοι μηχανισμοί για να υποβάλλονται καταγγελίες σε περίπτωση που δεν συμμορφώνεται η χώρα με τις ε, οδηγίες. Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία έχει στόχο την αποφυγή ε, δημιουργία τέτοιων γκρίζων ζωνών. Στόχος είναι να βρούμε τρόπους έτσι ώστε αυτοί οι εργάτες να νομιμοποιηθούν και να μην είναι πλέον παράτυποι έτσι ώστε να έχουν το δικαίωμα στην εργασία. Διαφορετικά να επαναπροωθηθούν με ασφάλεια. Σε ό,τι αφορά τους ε, εργαζόμενους, η οδηγία για τους εργαζόμενους παρέχει σαφείς διατάξεις ε, και υποχρέωση ε, τα κράτη-μέλη να έχουν κυρώσει σε περίπτωση που διαπιστωθεί εκμετάλλευση των ε, εργατών και να υπάρχουν επίσης οι μηχανισμοί έτσι ώστε ο εργάτης να λάβει την αμοιβή που δικαιούται ακόμα και αν δεν βρίσκεται νόμιμα στην επικράτεια της Ένωσης. Αυτό ισχύει λοιπόν για όλους, νόμιμους και μη εργαζόμενους. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει τις τοπικές και περιφερειακές αρχές στην ε, Ιταλία αλλά και σε όλα τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να καταπολεμηθεί το φαινόμενο αυτό. Το ε, Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης, ΆΜΙΦ, χρησιμοποιείται και θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό στην Ιταλία. Ε, χρησιμοποιούνται επίσης τα διαρθρωτικά ε, ταμεία και το ε, Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή την κατάσταση στην Ιταλία και να παρακολουθεί την σωστή εφαρμογή της οδηγίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Αναμένουμε τη γραπτή σας απάντηση. Ο κύριος Μαριάς έχει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, θεωρούμε την αναφορά πάρα πολύ σημαντική και γι' αυτό όταν υπευλήθη γραπτό αίτημα από τον συνάδελφο τον κύριο Ζαριανόπουλο προς τους συντονιστές εγώ προσωπικά και το ECR υποστηρίξαμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε με την κατεπίγουσα διαδικασία, την οποία και ακολουθούμε. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που κάναμε, διότι αυτά που ακούσαμε από τους αναφέροντες ε, επιβεβαιώνουν τη σοβαρότητα και το κατεπήγον της αναφοράς. Έχουμε πει ότι στα κατεπήγοντα πρέπει να βγάλουμε αυτές που είναι πραγματικά επίγουσες και όχι γενικώ ε, όποια ε, αίτηση ε, αναφορά πρέπει να υπάρχει. Δεύτερον, μου κάνει εντύπωση ότι βλέπω Ιταλούς συναδέλφου, θα περίμενα να τους δω εδώ για να ακούσουμε τη δικιά του άποψη για το τι συμβαίνει στην Ιταλία, γιατί αυτοί έχουν μια καλύτερη εικόνα. Αλλά είδαμε τα πράγματα, είναι δεδομένο ότι μέσα από την οικονομική μετανάστευση και στην Ιταλία αλλά και στις άλλες χώρες δημιουργείται ένας εφεδρικός στρατός, τον οποίο κρατούν στην παρανομία, δεν του δίνουν το δικαίωμα να αποκτήσουν άδεια παραμονής και όποτε θέλουν τους αξιοποιούν για εργασία δίνοντάς τους χαμηλούς μισθούς και όποτε δεν τους θέλουν τους εκδιώκουν. Άρα λοιπόν εδώ είναι μια κατάσταση ιδιαίτερα σοβαρή στα θέματα των εργατών γης, σε ένα κομμάτι που αφορά την κοινή αγροτική πολιτική που πέφτουν δισεκατομμύρια και θεωρώ ότι πρέπει η αναφορά αυτή να μείνει ανοιχτή μια και λέτε να επισπεύσω, να μείνει ανοιχτή η αναφορά, να μπορούμε να παρακολουθήσουμε τι γίνεται στο θέμα αυτό, να υπάρξει επιστολή στην Ιταλική κυβέρνηση για να μας απαντήσει συγκεκριμένα και ενδεχόμενα και στην περιφέρεια την αρμόδια γιατί μπορεί εργασιακά θέματα με βάση τον Ιταλικό νόμο να ανήκουν και σε επίπεδο περιφέρειας επειδή έχουν διάφορες βαθμίδες. Άρα λοιπόν όλες οι αρμόδιες αρχές να λάβουν την επιστολή μας λέγοντάς τους ότι αυτή η κατάσταση που επικρατεί είναι απαράδεκτη και θα πρέπει να προχωρήσουν με βάση ε, τα ισχύοντα και με τις διεθνείς συνθήκες και με βάση τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Ε, αυτό θα κάνουμε. Κατευθείαν. We are Θα διατηρήσουμε την αναφορά ανοιχτή και θα αποστείλουμε επιστολή στην Ιταλική κυβέρνηση ότι έχουμε κάθε λόγο να τους ζητούμε εξηγήσει σχετικά με το θέμα. Θυμίζω ότι είναι ευρωπαϊκό έδαφος και όπως θύμισε ο κύριος Μαριάς είναι απαράδεκτη η κατάσταση. Το πώς μεταχειρίζονται τους ανθρώπους αυτούς που εργάζονται, που δουλεύουν τη γη τους και που έχουν φτάσει με τις καλύτερες προθέσεις. Λοιπόν, αυτό θα κάνουμε. Προχωρώ τώρα επιταχύνοντας κάπως, γιατί ακόμα μισή ώρα πίσω είμαστε σε σχέση με το πρόγραμμα. 189 και 240 ο κύριος Αντώνιο Λουίθι Μπάσκεθ Ντελγάδο είναι εδώ. Σα δίνω το λόγο για 3 με 4 λεπτά παρακαλώ. Και όσο πιο σύντομα τόσο το καλύτερο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, Σα ευχαριστώ για το λόγο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ε, δυνατότητα αυτή και να μοιραστώ την ε, παρέμβασή μου με τον ε, εκπρόσωπο κύριο Εσπινόσα της οργάνωσης από τις ενώσεις δηλαδή αστυνομικών δυνάμεων σχετικά με την ισοτιμία των εισοδημάτων των μισθών τους και σε σχέση με τα όσα έκανε η κυβέρνηση και μιλούμε για μια διαδικασία που δεν ολοκληρώθηκε ή δεν συνέβη εχθές ή σήμερα, αλλά είναι 30 χρόνια που διαμορφώνεται. Εμείς ευχαριστούμε τις προσπάθειες όλων των μελών των υπηρεσιών επιβολής του νόμου στην Ισπανία, σε όλα τα επίπεδα, για τις προσπάθειες τους, λέγω, που είναι σημαντικές και προκειμένου να τις αξιοποιήσουμε θα πρέπει να διατηρήσουμε ανοιχτή την αναφορά αυτή γιατί άλλες τέσσερις συμφωνίες είχαν συναυθεί οι οποίες, τις οποίες αγνόησε παντελώς η Ισπανική κυβέρνηση. Ζητούμε λοιπόν να διατηρηθεί ανοιχτή η αναφορά γιατί έχουμε συγκεκριμένες ε, ε, υποβολές στα ε, επιμέρους κοινοβούλια, τα αυτονομικά κοινοβούλια, τις αυτονομικές κυβερνήσεις και την τελευταία φορά 13 Νοεμβρίου 316 βουλευτές υπερψήφισαν η πλειοψηφία του Εθνικού Κοινοβουλίου για την ε, ισοτιμία την μισθολογική, για την γεφύρωση του χάσματος του μισθολογικού μεταξύ των κεντρικών ομοσπονδιακών, αν θέλετε, να το πούμε έτσι, αστυνομικών δυνάμεων και των ε, αστυνομικών δυνάμεων των υπαλλήλων, δηλαδή των δυνάμεων των ε, αυτονομικών περιφερειών. Θα δώσω τώρα το λόγο στους ε, διοργανωτές αυτής της προσπάθειας και της αναφοράς αυτής. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα ήθελα να ευχαριστήσω για την προσοχή σας και την δυνατότητα που μας δίνετε για να παρουσιάσουμε την αναφορά αυτή σήμερα εδώ στο Κοινοβούλιο. Το μισθολογικό χάσμα των αστυνομικών δυνάμεων, των κρατικών και της Guardia Civil σε σχέση με τις ε, περιφερειακές αστυνομικές δυνάμεις της Καταλωνίας, της Ναβάρα και του Παΐς Βάσκο είναι στις συντάξεις, στα επιδόματα και στα συμπληρωματικά επιδόματα ε, τα μισθολογικά συνολικά σε πέντε επίπεδα. Είναι 30 χρόνια που συνεχίζεται αυτή η ανισότητα, αυτή η άνηση μεταχείριση μεταξύ των αστυνομικών δυνάμεων και που οι αυτονομικές ε, υπηρεσίες επιβολής του νόμου ζητούν να γεβηρωθεί 30 χρόνια και εδώ έχω μαζί μου από το 94 από την Βουλή στην Ισπανία αναφερόμαστε στην συμφωνία που είχε υπογραφεί το 1992 και το οποίο δεν είχε γίνει σεβαστό, δεν είχε συμμορφωθεί η Ισπανική κυβέρνηση ήδη από τότε. 24 χρόνια από εκείνη την ημερομηνία έχουμε μια ένωση ε, κοινωνίας των πολιτών όπου να ζητούμε ένα πλήρες ε, νομοθετικό πλαίσιο στο οποίο να υπάρχει επιτέλους μια μισολογική ισότητα μεταξύ των αστυνομικών υπαλλήλων. Σε 1,5 μήνα ε, συγκεντρώσαμε ένα αριθμό ρεκόρ ε, υπογραφών σχετικά με την πρωτοβουλία, αυτή τη λαϊκή πρωτοβουλία την νομοθετική, προκειμένου να εξισωθούν επιτέλους οι μισθολογικέ και συνταξιοδοτικές όπου έχουμε τεράστιες διαφορές της τάξης των 600 ευρώ και άνω και σε άλλες ε, κατηγορίες ε, μισθολογικές άνω των 1000, των χίλιων ευρώ ε, μισθολογικό χάσμα. Κατά τη διάρκεια των 30 αυτών ετών δεν συμμορφώνεται η Ισπανική κυβέρνηση. Εμείς ζητούμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να γίνει επιτέλους αυτό. Ζητούμε να λυθεί υπόψη η αναφορά μας και, και ζητούμε να παραμείνει ανοιχτή μέχρι να επιληθεί αυτή η άνηση μεταχείριση. Ζητούμε επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σημειώσει αυτή την άνηση μεταχείριση και να την μεταχειριστεί όπως μεταχειρίζεται άλλες περιπτώσεις άδικης κοινωνικής συμπεριφοράς. Αυτό ήδη το ανεγνώρισαν 316 βουλευτές μέλη της Ισπανικής Βουλής. Σας ευχαριστώ πολύ. Thanks to both of you. Ευχαριστώ και τους δυο σας. Είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λέτε. Το 16% είναι ο μέσος όρος για το μισθολογικό κενό για τους αστυνομικούς, τους γιατρούς, τους ε, δικηγόρους σε όλη την Ευρώπη και είναι ντροπή πραγματικά και μπράβο σας που το αναφέρατε. Θα καλέσω τώρα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, πάρει το λόγο. Ο Στέφαν Ούρσο, Σουηδός είστε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, δίκιο έχετε, σου ειδώσουμε. Ακούσαμε μεγάλη προσοχή τους αναφέροντες, διαβάσαμε φυσικά και την αναφορά και ενώ φυσικά κατανοούμε απόλυτα το τι σημαίνει να υφίσταται κάποιος διακρίσεις, να αισθάνεται πως αδικείτε Να ξέρετε ότι στις συνθήκες αναφέρονται οι διακρίσεις ε, βάση ε, του φίλου και άλλες περιπτώσεις διακρίσεων. Εσείς όμως αυτό που εστιάζετε είναι στο ότι δεν υπάρχει ίση αμοιβή για ίση εργασία. Και στο άρθρο 153 της συνθήκης δυστυχώς ε, δεν ε, ε είναι σαφή τα πράγματα, δεν έχουμε εμείς δυνατότητα να αντιδράσουμε. Ζητάτε δράση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν δεν κάνω λάθος, και δεν μπορούμε να αντιδράσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχετε και τον κύριο Κόρτα Ροντρίγκε μαζί σα. Θα θέλατε, κύριε Κόρτα Ροντρίγκε, να σχολιάσετε. Όχι. Ωραία, για την άλλη αναφορά. Ε, την 189. Έχετε κάτι να προσθέσετε. Ε, νομίζω όμω ότι δεν υπάρχει κάτι παραπάνω. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Τώρα, σε ό,τι αφορά την άλλη αναφορά, διαφέρουν λίγο τα πράγματα, διότι εδώ πρόκειται για διάκριση ε, ανδρών και γυναικών και πρέπει να γίνει ένα διαχωρισμό διακρίσεις ε, με αφορμή το φύλλο, δηλαδή δεν υπάρχει ίση αμοιβή ε, για ίση εργασία και μισθολογικό χάσμα. Αυτό είναι ένα πιο σύνθετο ζήτημα. Πολλοί είναι οι παράγοντες που το επηρεάζουν, η πολιτική, η αγορά, οι διακρίσεις εκεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φυσικά προσπαθεί να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα και τις δύο αυτές ε, προκλήσεις. Σας ευχαριστώ. Ακούσαμε την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα θα δώσω το λόγο στα μέλη της Επιτροπής και να ακούσω τι θέλετε να κάνετε, πώς θέλετε να προχωρήσουμε για αυτά τα δύο θέματα. Μπέατρις. Θα είμαι γρήγορη. Είναι αλήθεια ότι οι αρχές της ισότητας και της μη διάκρισης είναι κεντρικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ίδια εργασία, ίδιο μισθό. Αυτή είναι μια αρχή, δεν χρειάζεται να την υπενθυμίσουμε. Αν μάλιστα αυτή η διάκριση γίνεται εξαιτία ε, φίλου, ε, φιλής ε, και λοιπά, είναι πιο γνωστό φαινόμενο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση που πρόκειται για διαφορά μεταξύ ενστόλων, είναι ακόμα πιο ακραίο φαινόμενο κάθε φορά που ένα εργαζόμενο πληρώνεται λιγότερο από έναν άλλο για την ίδια δουλειά, θα πρέπει αυτό να δικαιολογείται. Ένα κράτο δεν μπορεί να είναι αυθαίρετο προ αυτό. Παρ' όλα αυτά, είναι αυτό που κάνει το Ισπανικό κράτος εδώ και 30 χρόνια. Δεν υπάρχει κανένας ε, λόγος που να δικαιολογεί ότι ε, ένας ένστολος ε, της αστυνομίας πληρώνεται λιγότερο από κάποιον της χωροφυλακής όπου και αν αυτοί βρίσκονται στο κράτος. Ιδιαίτερα αν πρόκειται για την περιοχή της Βαρκελόνης που, όπου υπάρχει ένας ε, εθνικισμός που ενδεχομένως οδηγεί σε τέτοιου είδους διαφορές των μισθών. Ε, μια πρωτοβουλία των πολιτών για αυτό το θέμα υποστηρίχθηκε από 500.000 άτομα από όλε τις πολιτικές ομάδες, εκτός βέβαια αυτών που προσπαθούν να δημιουργήσουν διαφορές και διάκριση μεταξύ των πολιτών. Θέλω να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθήσει το θέμα από κοντά και να αναλάβει δράση. Πρέπει να παραμείνει θεματοφυλάκα των συνθήκων. Επίσης, ζητώ να στείλουμε μια επιστολή στην Ισπανική Βουλή έτσι ώστε, στην, έτσι ώστε η Ισπανική νομοθεσία να ευθυγραμμιστεί ε, με την Ευρωπαϊκή και να παραμείνει ανοιχτή αναφορά μέχρι ότου υιοθετηθεί αυτός ο καινούριο νόμος ο οποίος ε, θα ε, εξαφανίζει αυτές τις διακρίσεις. Επίσης να πω ότι η αστυνομία και η χωροφυλακή ε, ε, ε, είναι όχι μόνο εξασφαλίζουν την ασφαλεία μας, αλλά καταπολεμούν την τρομοκρατία, τη διαφθορά και προστατεύουν το κράτος δικαίου και το σύνταγμα. Γι' αυτό τους χρωστάμε. Και αυτή η πρωτοβουλία της Χουσαπόλ, του Συνδικάτου των Αστυνομικών, αξίζει την προσοχή μας. Πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη. Ευχαριστώ. Είπα ένα λεπτό, ήταν τρία. Ο κ. Νάρτ, όταν οι διακρίσεις γίνονται για λόγους ε, ε φύλου, διαφοράς ε, φύλου, όλοι θεωρούν ότι είναι διάκριση, ενώ όταν ε, γίνεται για μεταξύ ανδρών και ε, ε, ε, όταν γίνεται για, σε διαφορετικές κατηγορίες εργαζομένων δεν θεωρείται διάκριση. Εδώ πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι όχι απλώς κάνουν το ίδιο έργο, αυτοί που πληρώνονται λιγότερο ίσως κάνουν και πιο δύσκολο έργο. Αυτό δεν εκπλήσει κανέναν φαίνεται. Αν δούμε το κείμενο του, ΗΕ του, του το άρθρο 7, αναφέρει ότι ο μισθό θα πρέπει να είναι ίδιος για ίδια εργασία και χωρίς διακρίσεις. Έχουμε 316 βουλευτές που για πρώτη φορά, μεταξύ αυτών σοσιαλιστές και το Λαϊκό Κόμμα, από το 92 σοσιαλιστές το ζητούν, το Λαϊκό Κόμμα που επίσης δεν έχουν διορθώσει την κατάσταση, τώρα λένε ότι θα τη διορθώσουν. Ε, στα, στην Ισπανία λέμε τα λόγια πετάνε, οι πράξεις μένουν. Ε, τώρα δεν ξέρω αν χαρακτηρίζονται από υποκρισία οι βουλευτέ αυτοί, αλλά τέλο πάντων εμεί πρέπει να στείλουμε μια επιστολή στην Βουλή, να του πούμε στο Ισπανικό Κοινοβούλιο, να πούμε ότι είμαστε, ανησυχούμε για αυτό το θέμα και να παραμείνει βέβαια ανοιχτή η αναφορά. Γιατί αλλιώ θα, θα γίνει αυτό που, που συμβαίνει από το 92, δηλαδή τίποτα. Πρόεδρο, ευχαριστώ πολύ. Κυρία Βαλίνα. Καταρχήν να ευχαριστήσουμε τους αναφέροντες για την παρουσία τους και για τις εξηγήσεις τους. Εξήγησαν πολύ καλά τα αιτήματά τους. Η αναφορά αυτή δεν αναφέρεται μόνο στο οικονομικό ή χρηματικό, αλλά μιλούν και για τα δικαιώματά τους, ε, υγείας, ε, απεργίας κλπ. Εμείς εδώ σε αυτήν την Επιτροπή Είμαστε συνηθισμένοι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι ασαφή στις απαντήσεις της ε, και να πετάει τον μπαλάκι αλλού. Οπότε δεν μας εκπλήσει και η τελευταία της παρέμβαση ε, περί απουσίας αρμοδιοτήτων. Απ' την άλλη μεριά είναι δύσκολο να γίνει η συνολική ανάλυση της κατάστασης των ε, ενστόλων και των σωμάτων ασφαλεία. Γιατί δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει πριν πάρουμε αποφασή να εξετάσουμε καλύτερο το θέμα. Αλλά το, αυτό που είναι σαφέ είναι ότι πρέπει να, δούμε πώ μπορούμε να εξασφαλίσουμε τα συλλογικά του δικαιώματα. Ε, καθήκον μα είναι να βελτιώσουμε και τι αδυναμίε που έχουν οι οδηγίε και οι κανονισμοί που υιοθετούμε. Συνεπώ. Ε, προτείνω η αναφορά να παραμείνει ανοιχτή και να γίνει μια μελέτη για την εργασιακή κατάσταση των εργαζομένων στα σώματα ασφαλείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Και σίγουρα να στείλουμε και μια επιστολή στην Επίτροπο Απασχόλησης για να ενδιαφερθεί για αυτό το θέμα. Uh, Ευχαριστώ, Σολεδά. Είστε η τελευταία ομιλήτρια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε τους αναφέροντες. Έχουμε δύο διαφορετικές αναφορές με δύο θέματα τα οποία έχουν σχέση με μισθολογικές διαφορές και διακρίσεις. Θα μιλήσω για τα σώματα ασφαλείας, αλλά θα πρέπει να αναφερθώ στην ανάγκη να εργαστούμε και νομοθετικά, σφαιρικά, προκειμένου να εξαφανιστούν αυτές οι μισθολογικές διαφορές. 16,5% είναι αυτή τη στιγμή η διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών. Είναι χρήματα τα οποία οι γυναίκες χαρίζουν στους άντρες. Τι μπορούμε να κάνουμε. Κομισιόν έχει πάρει μέτρα, αλλά δεν μπορώ να πω ότι είναι αποτελεσματικά. Συστάσεις, ένα πρόσφατο σχέδιο. Χρειαζόμαστε όμως μια οδηγία. που θα περιλαμβάνει τα διάφορες ε, συνθήκες που έχουν ε, υπογραφεί και την οδηγία του 2006 η συνεργασία για ίδια δουλειά, ή ίδιο μισθό για ίδια δουλειά. Σε ό,τι αφορά τα σώματα ασφαλείας, ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίασή τους. Δεν μπορώ να πω όμως ότι αυτή η διαφορά έχει σχέση με τον εθνικισμό. Χρειάζεται να αυξηθούν οι μισθοί, χρειάζεται να βελτιωθούν τα δικαιώματα. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα εθνικισμού. Ίσως ε, ε, δεν έχουν απλώς αναλάβει τις ευθύνες τους οι διάφορες κυβερνήσεις. 1,2 ε, δισεκατομμύρια ευρώ ε, είναι τα ποσά τα οποία έχει υποσχεθεί ο Υπουργό να δώσει μέχρι το 2020 για τα σώματα Ασφαλείας. Θα διεκδικήσουμε αυτά τα χρήματα και ελπίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί αυτό, αυτή η δαπάνη. Προφανώς να μην είναι ανοιχτή η αναφορά μέχρι ότου ο νόμος τον οποίο έχουν υποσχεθεί, έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση να υλοποιηθεί. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, προτείνω το εξής. Κρατάμε και τις δύο αυτές αναφορές ανοιχτές. Γράφουμε στις αρμόδιες εθνικές αρχές, υπενθυμίζοντάς τους το πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την μισθολογική διαφορά μεταξύ άνδρων και γυναικών. Αυτό για την ε, 189 ενώ για τη 240 θα κάνουμε το ίδιο, κρατάμε ανοιχτή την αναφορά και γράφουμε στις Ισπανικές αρχές, στην κυβέρνηση, για να αναφέρουμε, όπως είπατε και εσείς, ότι πρόκειται για την εθνική ασφάλεια, για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, για την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών και μιλούμε για δυνάμεις ε, εφαρμογής του νόμου Οπότε θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ε, νομίζω ότι συμφωνούν και οι αναφέροντες. Μπεατρής, ναι, συμφωνώ, αλλά πιστεύω θα πρέπει να αναφερθούμε ρητά στο ότι στηρίζουμε την υιοθέτηση της συγκεκριμένης νομοθεσίας ε, από την Ισπανία. Νομίζω ότι το νομοθετικό πλαίσιο θα δώσει μια λύση. Εμείς από εδώ δεν μπορούμε να τη δώσουμε χωρίς την αντίστοιχη νομοθετική δουλειά. Πρόεδρος, Ωραία, οπότε θα γράψουμε και στο Κοινοβούλιο. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Είστε αστυνομικοί και οι δύο. Ωραία. Νιώθω σαν να είμαι στο σπίτι μου. Ο, ο μπαμπάς μου ήταν ε, αστυνομικός. Α, είμαστε από τη χωροφυλακή. Όλοι εμείς, όλοι εσείς είστε από τη χωροφυλακή. Καταβλητικό, μπράβο σας. Ο πατέρας μου πέθανε πέρσι, θα ήταν περήφανος που έχω εδώ σε αυτή τη συνεδρία τόσους πολλούς αστυνομικούς. Ε, καλή επιστροφή. Λοιπόν, έχουμε τώρα άλλη μία αναφορά την 328 και πάλι επί της Συνομοσπονδίας Αστυνομικών Eurocop σχετικά με τα κοινωνικά δικαιώματα, το δικαίωμα απεργίας και το δικαίωμα στην υγεία και στην ασφάλεια των αστυνομικών. Η ε, κυρία Άντζελς Μπος Κομπρέθιος. Παρακαλώ. Τέσσερα λεπτά αν μπορείτε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλό απόγευμα σε όλους. Η Eurocop εκπροσωπεί μισό εκατομμύριο αστυνομικού στην Ευρώπη και υπέβαλε τρεις ε, διαφοροποιημένες αναφορές που η Επιτροπή αποφάσισε να ομαδοποιήσει σε μία σχετικά με το δικαίωμα απεργίας το οποίο σχετίζεται με τις συλλογικέ διαπραγματεύσεις και τα λοιπά κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα όπως ε, εκείνο της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας εργασίας. Το, η κάθε μία από τις ε, πτυχές αυτές έχει το δικό της νομοθετικό πλαίσιο, αλλά μιλούμε για αναγνωρισμένα κοινωνικά δικαιώματα και τα οποία ε, προκαλούν μεγάλες διαφοροποιήσεις με τα υπόλοιπα κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών. Υπό το άρθρο 2 της οδηγίας ε, έχουν οδηγηθεί τα, κράτα, τα κράτη-μέλη σε τελείως διαφορετική νομοθέτηση σχετικά με θέματα που αφορούν στην προστασία της υγείας. Ζητούμε μια ευρωπαϊκή ρύθμιση νομοθεσία όπως γίνεται για τους εργαζόμενους στη θάλασσα. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια ε, και μιλούμε για, για, για μέσα προστασίας πάρα πολύ απλά όπως γάντια ή ε, ε, κράνος ή τέτοια πράγματα. Ζητούμε λοιπόν μια συγκεκριμένη νομοθετική πρόβλεψη σχετικά με την προστασία των αστυνομικών απέναντι στους κινδύνους που μπορούν να είναι παρόντες στην εργασία τους. Η Κομισιόν δεν αναφέρει στο σημείο μου από απέστειλε ότι οι 89 656 σχετικά με την ελάχιστη, τον ελάχιστο εξοπλισμό ασφαλείας ε, εξαιρείται υπό το άρθρο 2. Δηλαδή οι αστυνομικοί καλούνται να τρέξουν προς τον κίνδυνο ενώ όλοι οι υπόλοιποι πολίτες πρέπει να απομακρύνονται γρήγορα από τον κίνδυνο. Και για τον λόγο αυτό θα πρέπει τουλάχιστον μια πρόσθετη συγκεκριμένη πρόβλεψη για την ασφάλεια των ανθρώπων αυτών, των αστυνομικών, να αναλάβουμε. Το οποίο σημαίνει, για παράδειγμα, να ρυθμίζουμε την κατάρτιση των συγκεκριμένων ομάδων, των ατυχημάτων στην εργασία, για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τους εργαζόμενους αυτούς. Είναι αρμοδιότητα και ευθύνη των κρατών μελών. Αποφεύγει, αποφεύγουμε να έχουμε μια οδηγία πλαίσιο αλλά αυτό θα μας προσέφερε να αποφύγουμε πάρα πολλά ατυχήματα ε, σχετικά μεταξύ άλλων με τη χρήση των αλεξίσφαιρων γυλαίκων. Όπως συνέβη δυστυχώς πριν από λιγότερο από ένα μήνα με την δολοφονία αστυνομικού στη Γρανάδα. Αρκετοί λοιπόν αστυνομικοί στις ευρωπαϊκές χώρες θα υφίστανται ακόμα διακριτική μεταχείριση και άνηση μεταχείριση και θα είναι εκτεθειμένοι στους κινδύνου της εργασίας τους λόγω της έλλειψης αυτού του εναρμονισμένου πλαισίου αυτής τη οδηγίας λέσιο. Χρειάζεται λοιπόν ρητή αναφορά ή στον εξοπλισμό της προσωπικής ασφάλειας των αστυνομικών και την αναγνώριση των ε, επαγγελματικών κινδύνων και ασθενειών που σχετίζονται με την ε, απασχόληση των ανθρώπων αυτών. Υπό το άρθρο 28 της ε, Χάρτας Ανθρωπίων Δικαιωμάτων δεν μπορεί να περιοριστεί σε καμία περίπτωση το δικαίωμα στην απεργία των αστυνομικών υπαλλήλων. Και η αρμόδια επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης τοποθετήθηκε σαφώς σχετικά με το 6-4 της Χάρτας των ε, Δικαιωμάτων της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τον περιορισμό του δικαιώματος απεργίας των αστυνομικών υπαλλήλων. Ακόμα και οι έκτακτοι υπάλληλοι έχουν δικαίωμα στην απεργία. Προφανώς όπως υπάρχει μια ε, ε, υπηρεσία επιγόντων περιστατικών στα νοσοκομεία. Αντίστοιχα μπορεί να υπάρχει και τέτοια υπηρεσία στις αστυνομικές υπηρεσίες, αλλά υπάρχει ε, αλληλουχία ώστε να μην περιορίζεται το δικαίωμα των αστυνομικών εργαζομένων ή στην απεργία ή στις συγκεντρώσεις ή στην ενημέρωση τη συνδικαλιστική, στις συλλογικέ διαπραγματεύσεις. Αυτά είναι δικαιώματα τα οποία περιορίζονται και βάλλονται συστηματικά μεταξύ των υπαλλήλων των αστυνομικών δυνάμεων στην Πορτογαλία, στην Ιρλανδία ή στην Ισπανία. Όπως και στο παράδειγμα της Καταλόνιας, όπου, όπου αρνείται συστηματικά η κυβέρνηση το, την, το δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσης των αστυνομικών υπαλλήλων. Πρέπει να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των υπαλλήλων αυτών αντίστοιχα με εκείνο των δικαστικών ε, λειτουργών ή των πυροσβεστών και άλλων σωμάτων ε, για την ασφάλεια του κοινού. Η Κομισιόν λοιπόν απλώς μας αποστέλει μια, ένα σημείωμα που λέγει ότι πρέπει να συνεχίσουμε να επιτρέπουμε τις ε, αποκλήσεις αυτές μεταξύ κρατών μελών τις νομοθετικές και οι οποίε αφορούν σε θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και εργασιακά δικαιώματα που θα επιτρέπουν τη συνέχιση τη διάκριση μεταξύ των πολινών ανάλογα με το ποια είναι η χώρα στην οποία κατοικούν και ποιο είναι το επάγγελμα που εξασκούν. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ, λέει η Πρόεδρο. Σα ευχαριστώ πολύ που μα ενημερώσατε. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Σίλβη Φίν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να απαντήσει. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ως προς τα δικαιώματα των πολιτών, όλοι οι πολίτες είναι ίσοι όπως γνωρίζετε στο δικαίωμα στην πρόσβαση στην ασφάλεια, στα εργασιακά τους δικαιώματα, στο δικαίωμα στην απεργία, υπό την συνθήκη της Ένωσης. Για τις διατάξεις ή, ή στην υγεία στον χώρο αποσχόλησης, τα δικαιώματα των αστυνομικών υπαλλήλων καλύπτονται υπό κανονικές συνθήκες από τη διατάξη Ευρωπαϊκή Ένωσης Υγείας και Ασφάλειας που ισχύουν για τους αστυνομικούς υπαλλήλους όπως ακριβώς ισχύουν για τους υπόλοιπους εργαζομένους. Αυτό ακριβώς βρίσκουμε υπό την οδηγία πλαίσιο, αλλά βεβαίως υπογραμμίσατε και εσείς ίδια και εξηγείτε και στα έγγραφα που διανύματε, είναι ο εργοδότης που πρέπει να προχωρήσει στην ανάλυση κινδύνου. Επομένως, από τα κράτη-μέλη εξαρτάται να εφαρμόσουν την ορακή νομοθεσία. Υπάρχει μία εξαίρεση μειοψηφία λόγω της ιδιαίτερης φύσεως κάποιων συγκεκριμένων καθηκόντων ή στην άσκηση των καθηκόντων τους, δηλαδή της αποτελεσματικής προστασίας της κοινωνίας, προβλέπει η οδηγία πλαίσιο οι υποκανονικές συνθήκες να μπορούν να, αποσύρονται από μια εξαιρεση μειοψηφια λογω της ιδιαιτερης φυσεω καποιων συγκεκριμενων καθηκοντων η οποία θέτει σε κίνδυνο την ε, τη ζωή τους. Σε περιπτώσει όμως που όπως ρητά αναφέρει το νομοθέτημα θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή του, όπως έλεγα. Κατά τα λοιπά καλυπτόμαστε από τις διατάξεις της οδηγία Λέσιο και των λοιπόν οδηγιών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει την πρόθεση να προτείνει ιδιαίτερη συγκεκριμένη νομοθεσία η διάταξη για τους αστυνομικού υπαλλήλου. για το δεύτερο σημείο στο οποίο αναφέρεσαι, για το δικαίωμα απεργίας. Και εδώ υπογραμμίζεται σωστά ότι η συνθήκη αποκλείει το πεδίο του δικαιώματος στην απεργία. Αυτή καλύπτει υπό το κεφάλαιο 6 των, της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και στο πλαίσιο αυτό είναι το Δικαστήριο των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που αναφέρεται σε περιορισμό του δικαιώματο αυτού για τους αστυνομικού υπαλλήλου, αναφερόμενο σε λόγους ασφαλεία και συγκεκριμένων συνθήκων στην άσκηση του επαγγέλματος των αστυνομικών. Άρα λοιπόν είναι τα κράτη-μέλη που έχουν το περιθώριο στη διάθεσή τους προκειμένου να ρυθμίσουν τα θέματα αυτά. Και για να μην μακρηγορήσω, λέει εκπρόσωπος Κομισιόν, είναι ξεκάθαρα υπέρ της προώθησης των δικαιωμάτων αυτών, ιδιαίτερα υπό τον κοινωνικό πυλώνα που ανακηρύξαμε το 2017 και ο οποίος αποτυπώνει τα δικαιώματα και προσπαθεί να προστατεύσει τα δικαιώματα του συνόλου των εργαζομένων σε όλους τους τομείς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχουν οι συνάδελφοι, τα μέλη της Επιτροπής και σας παρακαλώ μας μένει μία αναφορά να εξετάσουμε. Ένα λεπτό ο καθένας, όχι παραπάνω. Μπέατρης. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα χρησιμοποιήσω αυτό το λεπτό που μου δίνετε. Ήθελα να θυμίσω στην Κομισιόν ότι εδώ δεν μιλούμε για ένα οποιοδήποτε δικαστικό σώμα. Ε, δηλαδή φαίνεται η Κομισιόν μας δίνει απλώς ερμηνείες νομικών κειμένων και στην νομοθετική πρωτοβουλία έχει συγκεκριμένη αρμοδιότητα και ρόλο η Κομισιόν ή στην ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας. Και καλό θα ήταν να ξαναδείτε το πλαίσιο της δυνατότητας παρέμβασής σας και ανάληψη πρωτοβουλίας νομοθετικής. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να μείνει ανοιχτή η αναφορά διότι είναι ουσιαστικό το ζήτημα κρίσιμης σημασία και θα ήταν πολύ χρήσιμο να αποστείλουμε μια επιστολή ή στα κράτη-μέλη που δεν συμμορφούνται προ το άρθρο 11 της Χάρτας των Δικαιωμάτων και ε, το αντίστοιχο κεφάλαιο σχετικά με τα δικαιώματα απεργία και τα συνδικαλιστικά. Πρέπει να είμαστε πιο προδραστικοί προκειμένου να συντονίσουμε την δράση των κρατών μελών, ιδιαίτερα όταν όλο και περισσότερο προχωρούμε προ Ευρωπαϊκή Ένωση με κοινή πολιτική ασφαλεία. Σα ευχαριστώ κύριο Μαριά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θεωρώ σημαντική την αναφορά. ευχαριστήσω την κυρία Άγγελς και την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία αστυνομία, την EuroCup, διότι τα θέματα που έθεσε πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Εδώ έχουμε ένα λειτουργήμα το οποίο έχει λόγω της φύσης του άμεση σχέση με τον κίνδυνο και εκ των πραγμάτων, εάν δεν υπάρχει ο αναγκαίος εξοπλισμός τον οποίο θα τον χορηγήσει η πολιτεία, οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται εκτεθειμένοι σε αυξημένο κίνδυνο για την υγεία τους την ώρα που ασκούν τα καθήκοντά τους. Αυτό είναι μια ιδιαιτερότητα και θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Αν δεν έχουν αλεξίσφαιρα γυλαίκα, εάν δεν έχουν τον εξοπλισμό τον κατάλληλο, εάν εκτίθεται συνεχώς σε κινδύνους, αυτό δεν αφορά μόνο την υγεία τους αφορά και τον τρόπο και τον χώρο εργασίας. Εδώ είναι λοιπόν κάτι το διαφορετικό. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι πρέπει να ληφθούν αυξημένα μέτρα σε σχέση με τον εξοπλισμό που πρέπει να παρέχει η πολιτεία για να δημιουργήσει τις συνθήκες εκείνες προκειμένου να εκτελούν τα καθήκοντά τους που είναι πάρα πολύ σημαντικά και για τη δικιά μας ασφάλεια κατά τρόπο που να μην εκτίθεται σε κίνδυνο η ίδια τους η υγεία, η ίδια τους η ζωή. Αυτό το στοιχείο, αυτή την ιδιαιτερότητα σε σχέση με την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των αστυνομικών πρέπει να τη δούμε με ιδιαίτερο τρόπο. Και γι' αυτό πιστεύω να μείνει ανοιχτή η αναφορά και να έχουμε συγκεκριμένα μέτρα για τη στήριξη των ετοιμάτων της Ευρωπαϊκής, Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Αστυνομίας που αυτά που είπε εφαρμόζονται πολύ περισσότερο για την Ελλάδα όπου δεν έχουν ούτε, αστυνο... ούτε γυλαίκα αλεξίσφαιρα ούτε τον εξοπλισμό η ελληνική αστυνομία και πρέπει να πάρει αυτόν τον εξοπλισμό για την ασφάλεια των αστυνομικών. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Νάρτ, που είναι πάντα επί του θέματος. Ε, πρόεδρε, δεν μπορεί να... <laughs> Δεν να έχουμε ποτέ, μάλλον υπάρχουν δύο πράγματα που δεν υπάρχουν καμιά αμφιβολία για αυτά. Είναι η βροχή στη θάλασσα, λέει ο μιλητή, και η απαντήση κομισιών. Αυτό που είναι απολύτω προφανέ είναι ότι μιλούμε για ένα θέμα που σημαίνει εναρμόνιση ζητημάτων ασφαλεία στην χώρο απασχόληση και στην περίπτωση αυτή το διακύβευμα είναι η ζωή των ανθρώπων. Των ανθρώπων αυτών προκειμένου να προστατεύσουν τη δική μα τη ζωή. Προκύπτει λοιπόν ότι όλα είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Επομένω, τελικά θα έχουμε την, την ένωση των κρατών που το κάθε κράτο κάνει ό,τι του κατέβει και όχι μια πραγματική Ευρωπαϊκή Ένωση. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Ας συνοψίσουμε λοιπόν. Θα κάνω κάτι που δεν έχω ξανακάνει μέχρι τώρα. Υπάρχει ένας Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και ε, την Υγεία στον χώρο εργασία στην Ευρώπη. Θα μπορούσαμε να του στείλουμε μία επιστολή όπου θα επισημένονται τα προβλήματα που ε, τονίστηκαν από την Συνομοσπονδία Αστυνομικών να τους καλέσουμε και να τους ε, παράσχουμε λοιπόν όλες τις ε, πληροφορίες. Από τη μία πρέπει να συμφωνήσουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ο έλεγχος και για την επιβολή της ε, νομοθεσίας και την εφαρμογή της οδηγίας είναι εθνική αρμοδιότητα. Εμείς μπορούμε να τους πούμε να το κάνουν, όμως αν τα κράτη-μέλη δεν εφαρμόσουν την οδηγία δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό μπορούμε να κάνουμε λοιπόν στην περίπτωση αυτή και νομίζω πως ε, πρώτη φορά στην Επιτροπή Αναφορών, όσο είμαι εγώ πρόεδρος τουλάχιστον, ε, θα ε, δώσουμε τη δυνατότητα σε αυτόν τον οργανισμό να συμμετάσχει στο έργο μας. Ας δώσουμε μια προθεσμία, ας πούμε, έξι μηνών και μετά θα προβούμε σε αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Συμφωνείτε? Νομίζω πως συμφωνείτε όλοι, ακόμα και οι αστυνομικοί φαίνονται ικανοποιημένοι από την απάντηση αυτή. Excellent. And every... Πάρα πολύ ωραία. Όλοι είναι ικανοποιημένοι. Ολοκληρώνουμε λοιπόν το θέμα αυτό και μας μένουν 9 λεπτά πριν σταματήσει η διερμηνία για να εξετάσουμε την τελευταία αναφορά και θα προσπαθήσουμε να είμαστε αποτελεσματικοί. Καλωσορίζω λοιπόν τον Μιγγέλ Βισέντε στην Επιτροπή Αναφορών για να μας παρουσιάσει την αναφορά 419-2018. Σας δίνω αμέσως το λόγο για 5 λεπτά. Maximum. Το πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Η συγκεκριμένη αναφορά έχει σχέση με τις συνθήκες εργασίας, τις οποίες ονομάζουμε κοινωνική ζούγκλα, στους φωνηπιακούς και παιδικούς σταθμούς που εξαρτώνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Λουξεμβούργο. Η κατάσταση ξεκινάει από το Μάιο του 2004, ε, όταν εισήχθη ε, στην Ευρωπαϊκή Δημόσια Διοίκηση ε, το καθεστώς του συμβασιούχου. Δεν προέκυψαν βελτιώσεις από τότε. Μιλάμε για ένα εκπαιδευτικό ε, που όμως έχουμε ε, που περιλαμβάνει ε, δημόσιους υπαλλήλου, τον οποίο το καθεστώς διέπεται από τις εθνικές συμβάσεις εθνικό δίκαιο δεν εξαρτώνται από την Κομισιόν έχουμε συμβασιούχους που είναι μια άλλη κατηγορία ανάλογα με το ποιο είναι ο εργοδότη ε, και αυτοί διακρίνονται σε υποκατηγορίε. Έχουμε προσωρινού υπαλλήλου. Προσωρινοί θα μου πείτε. Είναι προσωρινοί όμω που εργάζονται στην ίδια θέση για πολλά χρόνια. Πόσο προσωρινοί είναι αυτοί. Οι συνθήκε εργασία και αμοιβή αυτών των διαφορετικών κατηγοριών είναι πολύ διαφορετικέ. Τεράστιε θα έλεγα κιόλα διαφορέ καταλαβαίνετε τι, ποιο είναι το, ποια είναι η ατμόσφαιρα που δημιουργείται στους βεφονιπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Οι αναφέροντες θεωρούν ότι πρόκειται για ένα επάγγελμα προστατευόμενο στην, ε, στην νομοθεσία του Λουξεμβούργου. Ε, οπότε δεν επιτρέπονται αυτές οι διαφορές. Ορισμένοι από τους συμβασίουχους ε, διαπράττουν και κοινωνικό dumping, διότι οι μισθοί αυτών είναι χαμηλότεροι από τους από τους μισθούς, από τον κατώτατο μισθό ενός ειδικευμένου εργάτη που είναι 2.458 ευρώ το μήνα στο Λουξεμβούργο. Η προσωρινή, η οποία μάλιστα είναι μεγάλης διάρκειας, ε, εργάζονται εδώ και πολλά χρόνια ως προσωρινή, ε, καλύπτουν πάγιες ανάγκες. Ε, τα συμβόλαιά τους δεν αναφέρουν ποιον αντικαθιστούν. όταν λύγει μια σύμβαση ανανεώνεται χωρίς να τηρείται η απαραίτητη προθεσμία ανάμεσα δύο συμβάσεις, το απαραίτητο χρονικό διάστημα ανάμεσα δύο συμβάσεις, που είναι το 1 τρίτο του προηγούμενου συμβολέου. Η οδηγία 104 του 2008 για τους προσωρινά εργαζόμενους αναφέρει ότι η μεταχείριση θα πρέπει να είναι ίση και ε, ότι δεν είναι δυνατό να καλύπτουν πάγιες θέσεις. Σε ό,τι αφορά το πρώτο, τα δικαιώματά τους ε, και τις συνθήκες εργασίας τους, ε, δεν τήρηται η οδηγία. Ε, και ούτε τηρείται και η δεύτερη απέτηση περί πάγιων θέσεων. Ορισμένοι από τους ε, προσωρινούς υπαλλήλου ε, περνούν εξετάσεις για να γίνουν προσωρινοί, ε, για να γίνουν ε, συμβασιούχοι αλλά και πάλι το καθεστώ τους θα υπολείπεται έναντι των υπολείπων. Η κατάσταση είναι ε, σχεδόν κομική Σας ζητούμε να ζητήσετε, να ε, απαιτήσετε από την Κομισιόν να διορθωθεί αυτό, αυτή, αυτό το ιστορικό λάθος, να μην είναι ανοιχτή η αναφορά καθώς ο χρόνο ε, η διάκριση παραμένει και αν μου επιτρέπετε θα ήθελα να πω και το εξής. Μιλήσαμε για το κόστος ζωής στο Λουξεμβούργο, δευτερευόντως όμως, προκειμένου να υποδείξουμε, να αναδείξουμε το πρόβλημα. Αν θέλετε να ζητήσω από κάποιον από τους συνοδούς μου, ε, δεν, ε, δεν θα έχουμε χρόνο, πλέον κλείνει η διερμηνία, δεν θα έχουμε διερμηνία σε τρία λεπτά. Δυστυχώς πρέπει να σταματήσουμε εδώ για να ακούσουμε την Κομισιόν και τους συναδέλφους. Ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε. Όχι, όχι. Ήδη ξεπεράσατε τα πέντε λεπτά. Λυπάμαι. Πρέπει να περάσουμε το λόγο στην Κομισιόν. Αλλιώς δεν θα καταλάβετε τις ε, απαντήσεις. Κομισιόν. Δυστυχώς χωρίς μικρόφωνο. Ε, εκφράζω την άποψη της Κομισιόν, όχι του Κοινοβουλίου. Ας δούμε λίγο το ιστορικό αυτής της υπόθεσης από το 2004. Ε, είχαμε υπαλλήλους του δημόσιου υπαλλήλου ε, του Λουξεμβούργου. Ε, ορισμένες, από αυτούς προτάθηκε σύμβαση εργασίας, ορισμένοι τη δέχτηκαν, άλλοι παρέμειναν υπάλληλοι. Από τότε όμως δεν έχει γίνει κανενός είδους πρόσληψη με βάση την Εθνική Νομοθεσία του Λουξεμβούργου. Όσοι είχαν μείνει, ήταν προσωπική του επιλογή και γι' αυτό το λόγο μέχρι να συνταξιοδοτηθούν παραμένουν. Έχουμε πράγματι τρει κατηγορίε. Έχουμε δημόσιου υπαλλήλου του Λουξεμβούργου, έχουμε συμβασιούχου και έχουμε και προσωρινού υπαλλήλου. Σε ό,τι αφορά τον εξορθολογισμό τη κατάσταση. Χρειαζόμαστε προσωρινούς υπαλλήλου για λόγους γλωσσικούς. Έρχομαι, για παράδειγμα, κατά καιρού παιδιά τα οποία μιλούν γλώσσε οι οποίε δεν καλύπτονται από το διδακτικό προσωπικό. Και δεύτερον, ε, οργανώνουμε διαγωνισμού για συμβασιούχου, στου οποίου κάποιοι προσωρινοί πάλι λαμβάνουν μέρο. Και όταν τους περάσουν, γίνονται συμβασιούχοι οι συνθήκε είναι προφανώ ότι δεν είναι τόσο κακέ προκειμένου αφού τόσοι πολλοί προσωρινοί δέχονται να περάσουν το διαγωνισμό. Ευχαριστώ πολύ. Ποιο Μαρτά. Ένα λεπτό έχω στη διάθεσή μου. Θα προσπαθήσω να πω τα πιο σημαντικά. Έχω την εντύπωση ότι επαναλαμβάνομαι. Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τέτοιου είδου αναφορέ. Κατηγορούνται τα θεσμικά όργανα τα οποία προσπαθούν να κηρύττουν την αλήθεια σε οποιονδήποτε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά όταν πρόκειται για τον εαυτό τους ε, παραβαίνουν την νομοθεσία. Και εν πάση περιπτώσει, οποιαδήποτε και αν ήταν η επιλογή εκείνη τη στιγμή, το 2004, ε, δεν απαντάται για το θέμα των διακρίσεων. Δεν μας ενδιαφέρει το αν υπάρχουν διαφορετικά καθεστώτα. Το σημαντικό είναι να μην υπάρχουν διακρίσεις. Υπάρχει και νομολογία της, του Δικαστήριου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καλεί όλα τα κράτη-μέλη να ευθυγραμμιστούν με την νομοθεσία. Δεν μας θα δώσατε απάντηση Κομισιόν. Δεύτερον, λέτε ότι δεν μπορείτε να αντικαταστήσετε όλους τους προσωρινούς για, λόγους, για το λόγο ότι αλλάζει το γλωσσικό προφίλ των μαθητών κλπ. Δεν, υπάρχει, δεν έχει κομισιόν υποχρέωση να καταρτίζει το προσωπικό της αν, υπάρχει, αν υπάρχουν ελλείψεις σε συγκεκριμένες γλώσσες, θα πρέπει να γίνει κατάρτιση των, του προσωπικού και σε αυτές τις γλώσσες. Έτσι εξασφαλίζουμε ευελιξία. Το κοινοβούλιο δε έχει καταδικαστεί επανειλημμένος για τον ίδιο λόγο ως διαχειριστής παιδικών σταθμών. Από ό,τι φαίνεται η Κομισιόν, ε, όπως κάνει και με, την, ε, τα δημοσιονομικά, έτσι και εδώ κάνει περικοπές ε, στους ε, μισθούς και επιβάλλει μια λιτότητα. Είναι, πρόκειται για παράνομες πρακτικές. Ευχαριστώ. Η διερμηνία ε, δυστυχώς εδώ πρέπει να διακοπεί. Ευχαριστώ Well, it's you